Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα αρχίζει ο πρώτος γύρος από τους συντονιστές. Ο Βέιν Φαμτεκάμπ από το ΕΛΚΑ έχει το λόγο πρώτος. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Την Τρίτη το βράδυ, στις 30 Σεπτεμβρίου, Είχαμε μια καλή ακρόαση με τον υποψήφιο επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς και την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή την Τετάρτη το επόμενο πρωί, στην Επιτροπή Μεταφορών ψηφίσαμε ομόφωνα για την έγκριση του κυρίου Σεύκοβιτς και πιστεύω πως μιλώ για όλη την Επιτροπή Μεταφορών. Η εμπιστοσύνη που δείξαμε στον Επίτροπο Σεύκοβιτς είναι παραμένει μεγάλη. Δεν θα συζητήσω τώρα τις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα και οδήγησαν στην αλλαγή χαρτοφυλακίου του κυρίου Σεύκοβιτς. Θα συνεισφέρει φυσικά πάρα πολύ στην Επιτροπή Γιούγκερ αυτό. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης της ε, Σλοβενίας δεν είναι και η καλύτερη, όμως δεν φταίτε εσείς γι' αυτό κυρία Μπούλτς. Διότι σήμερα έχουμε συναντηθεί για να εκτιμήσουμε τις ε, πολιτικές σας ικανότητες και στο μέτρο του δυνατού τη γνώση σας για το χαρτοφυλάκιο των ε, μεταφορών, το οποίο μελετάτε τις τελευταίες πέντε ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω θερμότατα εκ μέρους του ΕΛΚ. Δέκα συνάδελφους έχω, οι οποίοι θα σας κάνουν ερωτήσεις για τα διαφορετικά θέματα και οι ερωτήσεις αυτές θα είναι δίκαιες. Όπως είπατε και εσείς, χωρίς τις μεταφορές δεν κινείται τίποτα και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ευρωπαϊκή οικονομία. Και έχω λοιπόν τις ακόλουθες ερωτήσεις. Ο δικός χάρτης για, την, για τον ενίο χώρο ευρωπαϊκών μεταφορών. Τι θα κάνετε γι' αυτό, θα επιταχύνετε την εφαρμογή του, θα λάβετε υπόψη ε, τα όσα έχουν αποφασιστεί. Έπειτα, η χρηματοδότηση των ε, project 10T ε, και της διευκολύνσης ιδέωτας στην Ευρώπη. Από όσο ξέρω, το Συμβούλιο προσπαθεί να σπαταλήσει τα κονδύλια που διατίθενται για αυτά τα project. Και μας είπατε για τα 300 δισεκατομμύρια που σκοπεύει να διαθέσει ο κύριος Γιούγκερ. Φοβούμαστε ότι οι μεταφορές θα πάρουν την τελευταία θέση των προτεραιοτήτων και τι σκοπεύετε να κάνετε για να το αποτρέψετε. Επίσης, τι ε, σκοπεύετε να κάνετε για την αστική κινητικότητα. Διότι αν δεν κάνω λάθος θα είστε επίσης υπεύθυνοι για τον τομέα αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Επίσης, ε, οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν και αυτοί φυσικά δικαίωμα στις μεταφορές και τις χρειάζονται. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούλς, έχετε σχεδόν τρία λεπτά για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στις τέσσερις ερωτήσεις παρότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Πρώτα απ' όλα η Λευκή Βίβλος πιστεύω ότι είναι απολύτως αναγκαίες ε, διότι δείχνουν το όραμα που έχουμε. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε τομέα όπως και στο τομέα των μεταφορών χρειάζεται ένα τρόπο ώστε να ε, καταλάβει με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει. Αυτή είναι η χρησιμότητα της Λευκής Βίβλου. Κατά τη γνώμη μου δίνεται μια ε, κατεύθυνση, σωστή κατεύθυνση για το μέλλον μέσα στη Λευκή Βίβλο. Δεν θα επιφέρω αλλαγές, ε, δεν συνιστά αυτοπροτεραιότητα για μένα. Ξέρουμε όμως ότι σημειώνονται νέες εξελίξεις καθημερινά θα το παρακολουθούμε εκ του συνεγγύς με το επιτέλειο μου. Εάν ε, συντρέξει λόγος ε, θα εισηγηθούμε αλλαγές μετά από τις αξιολογήσεις που θα κάνουμε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής μεταφοράς. Εγώ πιστεύω στην διαρκή επικοινωνία με αυτούς που συμμερίζονται το όραμά, μας, όραμά μας για το μέλλον. Ας περάσουμε τώρα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν πολύ απλό λόγο, διότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο συνεχές ε, δίκτυο για να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μας επιτρέπουν να έχουμε την ευφυή βιωσιμότητα, ε, την ευφυή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, την ευφυή βιωσιμότητα. Αυτό μας προσφέρουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα που προκύπτουν από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτού έχουμε και τον κατάλληλο μηχανισμό για να τα χρηματοδοτήσουμε. Πέρα από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς έχουμε και προτεραιότητες ε, τις οποίες έχουμε ιεραρχήσει για το μέλλον των διευρωπαϊκών δίκτυων. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες. Ας περάσω ε, στη τρίτη και τέταρτη ερώτηση. Αστική κινητικότητα. Πολύ σημαντικό αυτό Συμβαίνει όμως σε εθνικό επίπεδο. Εμείς από πλευράς μας θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε έναν συντονισμό, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη με κάποια μέτρα, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που θα έχουν οι εθνικές πολιτικές και να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Για τη συνεργασία Βλέπετε ποια είμαι, θα είμαστε σε διαρκή διάλογο όπως και με τους ε, συναδέλφους επιτρόπους. Σας ευχαριστούμε. Ισμελ Ερτούκ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Μπούλτς. Αναφέρατε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αναφέρατε σαφέστατα ότι εσείς δεν θα επιτρέψετε το κοινωνικό dumping και τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει τα πράγματα πάρα πολύ μονόπλευρα όσον αφορά την ε, απελευθέρωση. Γι' αυτό λοιπόν και θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε υποψήφια Επίτροπε, ποιοι είναι οι στόχοι ή τα μέτρα τα οποία θέλετε να εισαγάγετε έτσι ώστε να διασφαλίσετε τα κοινωνικά δικαιώματα και τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα μεταφορών και να τον βελτιώσετε. Και επί, ε, πλέον είστε έτοιμοι να εισαγάγετε στην ε, νομοθεσία κλαδικές συμβάσεις και σταθερές τιμές. Έπειτα, χρηματοδότηση των υποδομών. Αναφερθήκατε σε αυτές και αναφερθήκατε και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και στη διευκολύνση συνδέοντας την Ευρώπη. Προσπαθούμε λοιπόν να χτίσουμε ένα δίκτυο βασισμένο σε αυτά. Σε πολλές όμω χώρες υπάρχει μια συζήτηση για τα διόδια, Κυρίω στην δική μου την πατρίδα, στο, νότο της Γερμανίας. Έχετε συγκεκριμένους στόχου όσον αφορά την χρηματοδότηση για τις υποδομές σχετικά με ένα τέτοιο σύστημα διοδίων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Okay, Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω αυτό το ερώτημα που θέσατε για τα κοινωνικά δικαιώματα. Όπως έλεγα και στην επιστολή μου, Πιστεύω ότι συνιστά αυτό μεγάλο επίτευγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι κατοχυρώθηκαν αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα. Κάποιοι τα θεωρούν ε, κόλλημα. Θα πρέπει να μετατρέψουμε τα κοινωνικά ε, δικαιώματα σε πλεονέκτημα για τα επιχειρησιακά μοντέλα που εφαρμόζουμε στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, από κοινού μπορούμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο ε, ανάπτυξη, βιωσιμότητα, πλήρη συμμετοχή. Αυτή, αυτά είναι τα σλόγγαν της ευρωπαϊκής οικονομίας και καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι ε, διαφυλάτοντας τα κοινωνικά δικαιώματα. Ας γίνω πιο συγκεκριμένη. Υπάρχει μια σημαντική κείμενη νομοθεσία για τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν ξέρουμε όμως ποια κράτη-μέλη εφαρμόζουν τι και σε ποιο σημείο ε, βρισκόμαστε. Ε, μελετώντας τα σχετικά έγγραφα για να προετοιμάσω την ακρόαση, αυτό διαπίστωσα. Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να ξέρω ποιο κράτος μέλος έχει εφαρμόσει ποια νομοθετήματα, ούτω ώστε να αναλυφθούν κάποια απαραίτητα μέτρα για να υπάρξει πλήρης μεταγραφή στην εθνική νομοθεσία των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Στη συνέχεια, η κοινωνικού περιεχομένου νομοθεσία ε, πρέπει να συμπεριληφθεί στο περίφημο refit. Ε, δηλαδή, ε, μπορούμε να είμαστε απλούστεροι, να είμαστε σαφέστεροι σε σχέση με αυτά που θέλουμε να εφαρμοστούν, ούτως ώστε αυτοί που καλούνται να τα εφαρμόσουν να κατανοήσουν καλύτερα ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Σε όλους τους τομείς, στις οδικές, εναέρειες, σιδηροδρομικές, ε, ε, θαλάσσιες μεταφορές, σε όλους τους τομείς, ε, θέλω να είναι διαρκής ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς. Θα επιμείνω σε αυτό. Δεν είμαστε εχθροί. Εάν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, και αυτό μου δείχνει και η προσωπική μου εμπειρία, εάν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, σίγουρα μπορούμε να βρούμε λύσεις. Ε, αυτή θα είναι η στάση μου. Σίγουρα ε, ορισμένες φορές είναι δύσκολα τα πράγματα και φαίνονται ανεπίλητα τα προβλήματα. Παρόλα αυτά Πιστεύω ότι καλές λύσεις μπορούν να βρεθούν αν υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση εάν κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα ζητήματα. Κάτι άλλο που επίσης σχετίζεται με τα κοινωνικά δικαιώματα είναι αυτή, αυτό το χάσμα ανάμεσα στην απίστευτη πρόοδο κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές ε, και ε, το χάσμα λοιπόν με τον διωγγούμενο αριθμό των νέων ανέργων. Πιστεύω ότι μέρος της προσπάθειας ε, θα είναι να εξασφαλίσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και για τις γυναίκες να μπουν σε αυτό το κλάδο ο οποίος ε, σημειώνει μεγάλη πρόοδο από τη μία, από την άλλη είναι ιδιαίτερα υψηλή η ανεργία με τους ε, συναδέλφους ε, επιτρόπους που είναι αρμόδιοι, συναρμόδιοι μάλλον για αυτά τα ζητήματα, θα διαβουλευτώ τόσο ώστε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση από κενού. Υπάρχει και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να απαντήσω, το θέμα των διοδίων. ο ρηπαίνων πληρώνει, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο χρήστης πληρώνει. Είναι δύο βασικές αρχές. Φυσικά, σε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος δικαιούται να επιλέξει τους τρόπους με τους οποίους ε, χρηματοδοτεί την υποδομή. Γιατί η γερμανική αυτή υπόθεση, ε, ε, φήμες, έτσι έχω ακούσει, δεν, έχω, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα, θα πρέπει να είμαστε πιστοί στις ευρωπαϊκές αξίες. του τέστην απουσία διακριτικής μεταχείρισης που να απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Κράμε, ευχαριστώ. Ρόμπερτ Ζήλε από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη, κυρία Μπόλτς. Ταυτόχρονα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο γιούνκερ για την δομή που έχει δημιουργήσει. Δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα τα πράγματα. Ίσως ε, η Επιτροπή Μεταφορών θα έπρεπε να αποκληθεί επιτρο... πυροσβεστική υπηρεσία μεταφορών και πολιτικών προβλημάτων, ομάδα πυροσβεστών. Έτσι θα μπορούμε να βοηθούμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στη θέση αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ποια είναι η αντίδρασή σας στο τέλος του 2016 όταν θα είναι σαφές ότι κάποιο κομμάτι, κάποια τα προγράμματα της διασύνης της Ευρώπης που συνδέονται με τις χώρες συνοχής δεν θα έχουν προχωρήσει καθόλου. Πώς θα αντιδράσετε, πώς θα κινηθείτε να μην χαθούν πόροι, και να μην χαθούν οι επενδύσεις όσον αφορά τις μεταφορικές υποδομές όπως αναφέρατε στην εισαγωγική σας ομιλία απάντηση ευχαριστώ θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε μια έννοια που έχει αναφερθεί παλιά ή το χρησιμοποιήσει το χάνεις μεταφράζεται use it or lose it αυτή είναι σημαντική έννοια γιατί ήμουν υπουργό στη χώρα μου και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως της χώρας μου. Και αυτός ήταν το τομέας που έπρεπε να καλύψω. Και έβλεπα ότι υπήρχαν πολλές προκλήσεις, κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών. Τα κρίσιμα προγράμματα που ακολουθούν κρίσιμο μονοπάτι δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη αν τα ζωτικά προγράμματα δεν υλοποιούνται, δεν ολοκληρώνονται. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η έννοια χρησιμοποίησέ το ή θα χαθεί, καλή έννοια, διότι βοηθά εκείνους που έχουν επομιστεί ευθύνες να ολοκληρώσουν ένα έργο. Είναι πολύ καλό κίνητρο. Δεν σημαίνει όμως ότι οι χώρες θα χάσουν τα χρήματα. Τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται καλά από εκείνους που δεν έχουν υλοποιήσει σωστά τα προγράμματα ε, επιστρέφει στο κοινό ταμείο και από το ίδιο κοινό ταμείο ξαναπαίρνουν χρήματα οι χώρες για να τα ξαχρησιμοποιήσουν. Δεν χάνεται για τις χώρες το ποσό, αλλά συνεπιφέρει κάποια πειθαρχία. Κανείς δεν σπρώχνει τις χώρες να καθορίσουν ημερομηνίες. Οι χώρες αυτοβούλως καθορίζουν ημερομηνίες. Να σας πω και κάτι ενδιαφέρον. Μόλις ανέλαβα τα ταμεία συνοχής στη Σλοβενία, είδα ότι ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι είναι δικά του τα χρήματα. Το Ταμείο Συνοχή Σλοβενία είναι χρήματα τη Σλοβενία που τα παίρνουμε μέσω των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ενώση και έχουμε δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, πολλά κίνητρα μπορούμε να προβάλλουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις. Κυρίως στο επίπεδο των κρατών μελών. Θα αφοσιώσω πολλή ενέργεια στην επικοινωνία, να εξηγήσω ποιες είναι οι ευθύνες ποιων στο επίπεδο χώρας ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Μπόλτς για την απάντησή σας. Ήταν μακρά η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή και τι μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έννοια του εργαλείου Connecting Europe. Χρησιμοποιείται πόρη και από το Ταμείο Συνοχής, με τους κανόνες του Ταμείου Συνοχής για να δημιουργηθούν διάφορα προγράμματα ε, για διέλευση που συνδέει πολλά κράτη-μέλη. Και συζητάμε πάντα αυτή την περίπτωση. Αν κάποιος δεν είναι έτοιμος, δεν είναι τρία κράτη-μέλη, δεν έχουν έτοιμα τα προγράμματα, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθούν ε, τα χρήματα σωστά. Θα χρησιμοποιηθούν από τις χώρες που είναι πιο έτοιμες για άλλα προγράμματα, αλλά τις δεν τα χρησιμοποιούν. Α, διαφορετικά δεν θα υπάρχουν ε, δεν θα υπάρχουν πρόοδοι όσον αφορά τα προγράμματα του διαδρόμου. Φέρετε την ειλικρινή απάντηση. Θα θέλετε να απαντήσετε? Όχι τότε. Η Γκεζίνε Μάισνερ έχει το λόγο για την επόμενη ερώτηση εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και από εμάς τους φιλελεύθερους κύριε Μπούλτς. Αναφέρατε ότι για εσάς είναι πάρα πολύ σημαντική μια ενιαία αγορά μεταφορών στην Ευρώπη και αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε και εμείς σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και τελευταία υπήρχαν κάποια project τα οποία ανεξάρτητα από πολιτική ομάδα μας έβρισκαν όλους σύμφωνους οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και οι διευκολύνσει ιδέοντα στην Ευρώπη. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ αγαπητό σε εμάς, ιδιαίτερα σε μένα γιατί προέρχομαι από μια παράκτια περιοχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό επομένω να συνδεθούν όλα τα λιμάνια και εξωτερικά και εσωτερικά και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Για αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα να σας κάνω τις εξής ερωτήσεις. Καταρχάς όσον αφορά τους λιμένες, εσείς τι ε, φαντάζεστε πώς μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η ναυσιπλοεία στα λιμάνια και να γίνει πιο ε, περιβαλλοντικά φιλική. Πώς μπορούμε να το σπρώξουμε προς τα μπροστά αυτό. Έπειτα, δεύτερη ερώτηση, εσωτερικές επλωτές οδοί. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που χρησιμοποιούμε. Εσείς ποιες τεχνικές δυσκολίες έχετε εντοπίσει, τι θα μπορούσε να κάνει κανείς έτσι ώστε να ενισχυθεί η εσωτερική ναυσιπλοεία και να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον. Και τρίτη ερώτηση, είπατε ή γράψατε μάλλον ότι εγώ καθοδηγούμε από τις λύσεις και αυτές έχω στο νου μου. Τι λύση νομίζετε πώς χρειάζεται ο ευρωπαϊκός χώρος των ε, μεταφορών ε, λοιπόν και πώς μπορούμε να ε, τον εφαρμόσουμε και τι σχέση θα έχει αυτό και για τους ανθρώπους αλλά και για τις κυβερνήσεις που, για όλους δηλαδή που θα χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πιεστεί, τότε θα περιμένουμε πάρα πολύ για να γίνουν πράγματα. Εσείς λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε και τι θα θέλετε να γίνει έτσι ώστε να επισπευστεί η διαδικασία. Κυρία Μπούλτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρεις ε, σημαντικές ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τους λιμένες και με το πράσινο θεματολόγιο. Η δεύτερη για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Ε, καταρχάς, όσον αφορά τους λιμένες. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, οι λιμένες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Και η ναυτιλία είναι και η πιο κερδοφόρος επιχείρηση στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή σας είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και ακόμα πιο σημαντική. Πιστεύω πως έχουν γίνει αρκετά στον τομέα αυτό. Καταρχάς η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να μας βοηθά. Όχι μόνο ε, για τα πλοία και τις τεχνολογικές εξελίξεις, και να πω εδώ ότι μου έκανε τρομερά θετική έκπληξη όταν διάβασα ότι μερικά λιμάνια επιβραβεύουν τα πλοία που έχουν ε, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με χαμηλή φορολογία και πιστεύω πως είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Έπειτα άκουσα για, αυτά, για αυτές τις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πλοία αντί για καύσιμα όταν αράζουν σε ένα λιμάνι. Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική ενέργεια και αυτό είναι καταπληκτικό επίτευγμα πιστεύω όταν μιλάμε για πρασίνισμα και για πιο φιλικές ενέργειες προς το περιβάλλον. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για ναυτιλία και για πράσινο θεματολόγιο ε, πρέπει να συνυπολογίζουμε και την διάσταση των διεθνών συμφωνιών. Πρέπει δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε και τους ε, διεθνείς οργανισμούς, να τους ενημερώσουμε, να συνεχίσουμε την συζήτηση μαζί τους έτσι ώστε να ε, δρομολογήσουμε αυτήν την διεθνή συμφωνία για το πώς θα εφαρμόσουμε το θεματολόγιο αυτό. Αν δεν κάνω λάθος υπήρξε ήδη μια πρωτοβουλία για, κάποια με, ε, για κάποιους τρόπους μέτρησης του πρασινίσματος αυτού και για τρόπο μέτρηση για να δούμε αν ακολουθούνται αυτές οι περιβαλλοντικέ κατευθύνσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα και εγώ θα συνέχιζα να ενθαρρύνω αυτήν την εφαρμογή των πράσινων λύσεων και την σύνδεσή τους με τους λιμένες. Ας περάσω τώρα στην επόμενη ερώτηση για να προλάβω να απαντήσω σε όλες. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, που είναι επίσης πολύ σημαντική, είναι για τις εσωτερικέ πλειοτές οδού. Πιστεύω πως υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Σίγουρα δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη ε, τι ε, ίδιε δυνατότητε, όμως κάποια έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο δυναμικό για την εσωτερική ναυσιπλοεία και είναι πολύ σημαντικό να εξισωθούν αυτές οι εσωτερικές πλωτές οδοί με τους άλλους τρόπους μεταφοράς γιατί προς το παρόν ε, παρατηρείται ένας κατακαιρματισμός και οι περισσότερες ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό είναι μικρές επιχειρήσεις, πολλές φορές οικογενειακές. Ναϊάδες επίσης είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω πως μπορεί να βοηθήσει και σε επιχειρησιακό επίπεδο την ε, μείωση αυτού του κατακαιρματισμού, διότι διαφορετικά αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν από μόνες τους να βρουν μια ε, λύση διασύνδεσης κατάλληλη. Χρειάζεται σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας και χρειάζονται και κίνητρα και βελτιώσεις ως προς την τεχνολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μέρια Κίλονεν εκ μέρους της Γκουε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλετε να αποτρέψετε το κοινωνικό ντάμπινγκ στις ενιέρειες, εναέρειες, συγγνώμη, θαλάσσιες και οδικές μεταφορές. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Δεύτερον, η πολιτική μεταφορών είναι το μέλλον της Ευρώπης, διότι χρειαζόμαστε την ανάπτυξη. Η ψηφιακή προσέγγιση για την ε, επιμελητή και για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές έχει κέρια σημασία. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε αυτός ο τομέας να έχει σε παγκόσμιο επίπεδο ηγετικό ρόλο και οι υπηρεσίες να είναι διαλειτουργικές βιώσιμες και να προσανατολίζονται στον πελάτη. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε το υφιέστερο σε παγκόσμια κλίμακα ε, σύστημα μεταφορών. Πώς μπορούμε να δαπανίσουμε λιγότερα χρήματα και να έχουμε τα ε, μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. κυρία Βούλς. Το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ε, ας αρχίσω με την πρώτη σας ερώτηση. Σε όλους τους τομείς των μεταφορών προκύπτουν ζητήματα με το κοινωνικό ντάμπινγκ σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά. Θα ήθελα να ε, επιβεβαιώσω και πάλι ότι είμαι κατά του κοινωνικού dumping ε, στον τομέα των ε, μεταφορών ε, με φορτηγά, των μεταφορών, το dumping είναι διαφορετικό από ότι στον τομέα των εναέριων μεταφορών, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρόκειται για στρέβλωση της οικονομίας. Με την αύξηση των κυρώσεων δεν πρόκειται να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Καινοτόμες λύσεις χρειαζόμαστε. Πώς μπορούμε να οργανώσουμε την, τον τομέα ούτως ώστε να μην μπορεί πλέον να προκύψει αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν αλλάξουμε την οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζουμε το πρόβλημα, αν διαπιστώσουμε για ποιο λόγο ανακύπτει κοινωνικό ντάμπινγκ, αν εκριζώσουμε τις αιτίες του κοινωνικού ντάμπινγκ θα μπορούσαμε να βρούμε ικανοποιητικές λύσεις. Με ρωτήσατε επίσης με ποιο τρόπο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της ε, οικονομική ανάκαμψης ο τομέα των μεταφορών. Ξέρετε, ε, έχει γίνει σκληρή η δουλειά ήδη, θα μπορούσα εγώ να ε, έχω τα εύσημα αν θέλετε, αλλά δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρήματα χρειαζόμαστε για να αρχίσει ο σχεδιασμός των βασικών διαδρόμων των διευρωπαϊκών δικτύων. Όπως και ο προηγούμενος συνάδελφος ε, με απασχολούν και μένα τα ζητήματα της ε, ε, επιτόπιας συνεργασίας και του συνδυασμού με τα διαρθωτικά ταμεία παραδείγματο χάρη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι επιπρόσθετες επενδύσεις. Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια επαρκή υποστήριξη για αυτά τα προγράμματα. Σίγουρα θα είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή αν εγκριθεί από εσά την Τετάρτη ο τομέας των μεταφορών και μπορούμε να δούμε στο πακέτο ε, των 300 δις με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να γίνουν αποτελεσματικές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Αν να πω και κάτι άλλο γιατί δεν έλειξε ο χρόνος. Η τεχνολογία εξυπηρε... μας εξυπηρετεί. Αυτός είναι ο στόχος της. Τι έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια. Φοβερές εξελίξεις. Ε, στην, ε, πράσινη, στο πράσινο θεματολόγιο εάν χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογικές ε, εξελίξεις ε, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να προκύψει μια ομοιόμορφη ε, διαρκής διαχείριση του δικτύου. Αυτοί οι μηχανοδηγοί, παραδείγματο χάρη, έχουν ε, πέντε διαφορετικά συστήματα αυτή τη στιγμή και προκύπτουν ατυχήματα με το ICT και με το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης θα αποφευχθούν όλα αυτά και σταδιακά αν ακολουθήσουμε τις δεσμεύσεις που ήδη έχει εγκρίνει το Κοινοβουλίο μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και σταδιακά να φτιάξουμε νέες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, Κανμαντέλη, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ λοιπόν ε, διότι δεν είχαμε απάντηση από πλευρά του κ. Γιούνκερ. Το λέω και πολύ ισχυρά οι μεταφορές δεν θα είναι η μεταβλωτή προσαρμογή της ε, μελλοντική Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μεταφορές είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που αξίζει. Δεν πρέπει να παίζονται μουσικές καρέκλες με αυτό. Είναι, αφορά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι κυρία Μπίλτς. Λοιπόν, σας εύχομαι το καλώς ήρθατε σε αυτή την ε, επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ σύντομη. Διαπραγματευόμαστε το πακέτο για το κλίμα, την COP21, ε, που θα γίνει στο Παρίσι συνεδρίαση και λοιπόν μεταφορές έχουν τον τρίτο νεκομό του θεκεπιού. Είναι αποφασιστική σημασία η αλλαγή του κλίματος. Όμως δυστυχώς οι μεταφορές ε, δεν μπαίνουν με τα δύο πόδια στην πολιτική για το κλίμα. Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Πώς θα τα καταφέρετε ούτως ώστε κοινωνικές, υγειονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές να αντιμετωπιστούν πώς θα δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης για τη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα του 2015. Δεύτερη ερώτηση, το Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής ε, ε, το, τη γραμμή ε, Λιόν τωρινου περίπου αυτό το πρόγραμμα ε, είναι άχρηστο και κοστίζει περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ απλή η ερώτησή μου. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους προγράμματα όπως το περίμονο τούνελ για τον Άνω Ρήνο στα πλαίσια της προσπάθειας της σύνδεσης Ευρώπης χωρίς να γνωρίζει το πραγματικό κόστος, χωρίς να γνωρίζει την ισορροπία του προπολογισμού και την επίπτωση που έχουν όλα αυτά τα προγράμματα στο περιβάλλον. Danke sehr. Frau das uh, Κοιτάξτε, απάντηση. Μεγάλη πρόκληση το πράσινο θεματολόγιο με τους στόχους. Υγείται των προσπαθειών Ευρώπη στον κόσμο και νομίζω ότι έχουμε πάρει τα πράγματα πολύ στα σοβαρά και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Μ' αρέσει η φύση, ζω στη φύση και πραγματικά σέβομαι τη φύση και γνωρίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μεγάλο σεβασμό για αυτήν. Τι έκανε τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρώπη. Αυτά που έκανε ε, ίσως να μην ήταν αρκετά Ελπίζω συνεχώς να προσπαθούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Να πω ένα-δύο πράγματα που θεωρώ πολύ σημαντικά και συμπεριλαμβάνονται στο θεματολόγιο και στην στρατηγική για τις μεταφορές και πιστεύω ότι θα θρηστούν όλα αυτά τα στοιχεία και τελικά οι μεταφορές θα μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το πρασίνισμα της οικονομίας. Έχει προοδεύσει η τεχνολογία σε όλους τους τομείς και ανέφερα ένα-δύο πραγματικά παραδείγματα επ' αυτού. Μετά πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά του κόσμου και αλλάζει η συμπεριφορά και μπορούμε να πετύχουμε εκεί περισσότερα διότι η πίεση των καταναλωτών είναι η καλύτερη δυνατή. Είναι δύσκολο να δώσει κανείς κίνητες επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνω αυτό υπόψη με άλλα κίνητρα. Αν οι καταναλωτές όμως είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και αν επιβαρύνονται εκείνοι που ρηπαίνουν με το κόστος ρήπανσης, τότε πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων. Πιστεύω ότι η σύνολος Κορυφής των Παρισίων είναι μεγάλο κίνητρο. Πιθανότατα δεν θα είμαι εκεί, αλλά αν είμαι μέλος της ομάδας σχεδιάζω να καθίσω μαζί με τους επιτρόπους που θα πάνε εκεί και θα έχουν πιο άμεση ευθύνη για το πράσινο θεματολόγιο και θα είμαι πολύ συνεργάσιμη θα ετοιμάσουμε δηλαδή πάρα πολύ καλό υλικό, το οποίο θα αντιπροσωπεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ανέφερα τη συμπεριφορά του κόσμου και την τεχνολογία. Όμως αναφερθήκατε και στο μεγάλο πρόγραμμα αυτό που συζητείτε πολύ συχνά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής ραχοκοκαλιάς. Τεράστιο έργο. Το θέμα είναι μπορούμε να πληρώσουμε τέτοιου είδους προγράμματα. Αν αμφισβητήσουμε τους διαδρόμους, ποτέ δεν θα λειτουργήσει η σπονδυλική στήλη, η ραχοκοκαλιά. Να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να το κουβεντιάσουμε όλοι μαζί και να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει και το εξής από τη στιγμή που θα έχουμε τη ρεχοκοκαλιά τη σιδηροδρομική θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα φορτία από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Βασικός μας στόχος αυτός, πέρα βέβαια από την κάλυψη των αναγκών των επιβατών. Αυτά τα μεγάλα έργα δημιουργούν θέσεις εργασίας, δημιουργούν ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα. Να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να ενθαρρύνουμε τη σωστή προσέγγιση, να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τη φύση αυτά τα έργα και οι τοπικές κοινωνίες να συνεργάζονται μαζί μας και το έργο να είναι εποφελές όχι μόνο για το σύστημα, για τη ραχοκοκαλιά αλλά εποφελές και για τις ε, τοπικές ε, κοινότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στον δεύτερο γύρο. Εδώ το λόγο έχουν τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και πρώτος είναι ο κύριος Τίτερ Λέμπρεχτ Κόχ. Δεν ακούει αρκετά καλά η κυρία Μπούλτς, λέει.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 σας άκουγα καθαρά, αλλά τώρα δεν σας ακούω καλά. Πρέπει να καταλαβαίνετε τα πάντα, να είστε σε αυτή τη θέση. Όμως αυτό είναι η δεύτερη φορά που μας συμβαίνει. Θα το βρούμε όμως. So, jetzt testen wir nochmal, ob es jetzt die Übersetzung besser ist. Hören Sie es jetzt? No? A little bit, but it was really good before. Und jetzt? Auch nicht? Yeah, I can hear, but very Okay, be patient with me. I will try my best, but uh, ja. understand that it's. Ja, nein, aber das müssen wir erklären, dass Sie richtig verstehen. Also wenn wir alle Englisch sprechen, wäre es einfach. Θα ήταν πιο εύκολο να μιλούσαμε όλοι αγγλικά, όμως υπάρχουν πολλές γλώσσες και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διερμηνίας. Θα δούμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί, όσος χρόνος χρειαστεί. Well, They tried their best as well. Yeah. Μάλιστα. Ορισμένες φορές λοιπόν είναι ε, καλό να υπάρχει χρόνος. Θα δώσω λοιπόν ε, το λόγο στον Dieter Λεμπρεχτ Κοχ, αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Κάθετε πίσω σας. Αριστερά πίσω σας. Πίσω σας είμαι κυρία Μπούλς, μάλιστα. Κάθε χρόνο σημειώνονται 250.000 ατυχήματα στους δρόμους της ε, Ευρώπης και υπάρχει ένα πρόγραμμα από το 2014 μέχρι το 2020 το οποίο έχει συνολικά περιεκτικές ε, προτάσεις για ε, μείωση κατά το ίμιση των σοβαρών ατυχημάτων στην Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα μέτρα που εσείς σκοπεύετε να πάρετε έτσι ώστε να γίνει ο στόχος του μείωσης των ατυχημάτων ή δυνατόν στο μηδέν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά θλιβερό όταν συμβαίνει ένα τύχημα, είτε στους δρόμους είτε οπουδήποτε αλλού. Και πραγματικά παίρνω το στόχο της Ευρώπης για τη μείωση στο μηδέν των ατυχημάτων πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρω πως είναι μάλλον αδύνατο να επιτύχουμε ένα τέτοιο στόχο, όμως πρέπει να δώσουμε ε, τον καλύτερό μας σε αυτό έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω πως υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης και αντιμετώπισης, όμως τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να μας βοηθήσουν να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ένα από αυτά που κάνουμε είναι να βελτιώνουμε καταρχάς τα ίδια τα οχήματα, να καταρτίζουμε, να εκπαιδεύουμε τους χρήστες έτσι ώστε να γνωρίζουν καλύτερα την οδική κυκλοφορία. Πιστεύω πως η εκπαίδευση και η κατάρτιση λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Χρειαζόμαστε κατάρτιση και χρειάζεται να το θυμόμαστε αυτό. Έπειτα, καλύτερη τεχνολογία, βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών, διασυνοριακή και ε, εθνική. Καλύτερη νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς και πάρα πολλά πρόσθετα μέτρα τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο κρατών μελών που να βελτιώσουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, να βελτιωθεί η σηματοδότηση στις οδικές κυκλοφορίες. Πρέπει όμως πραγματικά να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια περίπου έχουμε καταφέρει να έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Και ξέρω πως ε, δεν είναι, έχουν όλες οι χώρες τα ίδια αποτελέσματα λόγω της διαφορετικής οικονομικής κατάστασης. Όμως πιστεύω πως χρειάζεται να γίνει μια ανάλυση και να δούμε ποιες μέθοδοι έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να τις βελτιώσουμε και επίσης να συνεργαζόμαστε στενά με όσους διαχειρίζονται την κυκλοφορία έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Ιζαμπέλα Ντεμόντι από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ και από την πλευρά μου κάποια ερώτηση για την ασφάλεια, γιατί πιστεύω ότι στο πρόγραμμα του Γιούγκερ στην πρόταση με διάφορε προτάσει στο θέμα τη ασφαλεία αόριστα μόνο αναφέρεται. Και εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω εν γέννη, γενικά πέρα από το θέμα τη οδική ασφάλεια, πώ θα αντιμετωπίσετε το θέμα τη ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κέντρα και στι αστικέ περιοχέ. Thank uh, Ευχαριστώ. Στην Ευρώπη η ασφάλεια είναι ο τελικός στόχος, σημαντικότατο ζήτημα. Λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη για να βελτιωθεί η ασφάλεια. Δημιουργήσαμε τρεις υπηρεσίες. οι οδικέ μεταφορές δεν έχουν συγκεκριμένη υπηρεσία. Η νομοθεσία, οι συμφωνίες εφαρμόζονται σωστά σύμφωνα στις υπηρεσίες. Ε, επίσης η πιστοποίηση λαμβάνεται υπόψη και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες μέσω των φορέων αυτών να αυξήσουν τη σημασία που έχουν. Έχουμε αυτές τις υπηρεσίες, μπορούμε να τις δώσουμε περισσότερα περιθώρια να κινηθούν. Έτσι τα, θα πρέπει τα μέτρα ασφαλείας να εφαρμόζονται σωστά. Τι παρατηρήσαμε. Ότι σε επίπεδο χωρών κάποιοι νόμοι δεν εφαρμόζονται σωστά. Και εάν δεν εφαρμόζονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει την εφαρμογή των συμπεφωνημένων μέτρων, είτε μέσω των υπηρεσιών, είτε μέσω προσφυγής στο δικαστήριο κατά κάποιων χωρών, ούτως ώστε να εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ασφαλείας. Κάτι άλλο. Όσον αφορά την έννοια της ασφαλείας, τη γενικότερη, πρέπει συνεχώς να επιδιώκουμε καλή διαχείριση της κυκλοφορίας, καλό έλεγχο των υποδομών. Είδαμε πολλές επιτυχημένες περιπτώσεις στις μεταφορές. Κυρίως αυτό που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και στους σιδηροδρόμους. Ήδη έχει συμφωνηθεί το θεματολόγιο, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει ενιαίο σύστημα κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων. Και το σύστημα αυτό έχει συμβάλει στη βελτίωση της σημαντικής ασφαλείας των σιδηροδρόμων. Κάθε τομέας έχει δικά του θέματα. Προτεραιότητά μας όμως είναι να έχουμε σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας με σωστά συστήματα να είναι σαφέστατη η νομοθεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες να μας βοηθούν να εφαρμόζονται οι νόμοι σε τοπικό επίπεδο. Πέραν αυτού πρέπει να διερευνήσουμε το πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τα μέτρα ασφαλείας και οι επιβάτες και από πλευράς εκείνων που παρέχουν τις υπηρεσίες να το καταλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Μαριάν Τζαν Μαρινέσκου από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Στη Ρώμη θα στις αρχές Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών, έτσι ώστε να συζητηθεί ο νέος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν επιφυλάξεις για αυτό το πρόγραμμα. Εσείς τι άποψη έχετε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό project και εάν φτάσει ο χρόνος θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε τι στάση θα κρατήσετε εάν ένα κράτος ε, μέλος επιθυμεί και προτείνει αλλαγή για, τους, ε, για τις ευρωπαϊκές ε, διόδους. Απάντηση. Πιστεύω πως ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι ένα καταπληκτικό έργο. Και αυτό και από α, επιχειρηματική άποψη και από πολιτική, διότι αυτό που κάνει είναι από τη μία να βελτιώνει την κυκλοφορία, να βελτιώνει τη, τις οδούς και, εδώ θα ήθελα να απαντήσω στην τελευταία ερώτησή σας, διότι ήταν και μέρος της εναρκτήριας ομιλίας μου. Ναι, πιστεύω πως πρέπει να απλουστεύσουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν όντως κάποιες προκλήσεις σε ορισμένες χώρες επειδή έχουν κάποιες προστατευμένες περιοχές, όμως πιστεύω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο και να φροντίσουμε οι δύο δι αυτοί και οι άξονες κυκλοφορίας να είναι όσο το δυνατόν συντομότεροι, γιατί αυτό θα διευκολύνει και την κυκλοφορία. Τώρα, Όσον αφορά το ΣΥΣ2 και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, νομίζω αν δεν κάνω λάθος FAB λέγεται αυτό, και την διαχείριση των ε, σλό, των ε, χρονοθυρίδων, πιστεύω πως αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι βελτιώνει την διαχείριση των ε, οδών κυκλοφορίας και επίσης ε, μειώνει την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, ναι, φυσικά και θα προσπαθώ να βρώσω το δυνατόν περισσότερες λύσεις και να εξετάζω περισσότερες επιλογές. Πιστεύω πως ε, το project αυτό είναι καλό και χρειάζεται να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι σε αυτό και σε επίπεδο κρατών μελών φυσικά έτσι ώστε να ενοποιήσουμε την διαχείριση της κυκλοφορίας και να γίνει μια, η πλατφόρμα. Το λόγο έχει η Άννα Κλόντια Ταπαρτέλ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι κύριε Υποψήφια Επιτρόπε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η ερώτηση που έχω να σας κάνω έχει να κάνει με τα εξή θέματα. Η αύξηση της αστικοποίησης και η προσέλευση των ε, ανθρώπων στις ε, πόλεις έχει οδηγήσει στη ρήπανση και του αέρα αλλά και στην αύξηση της συγχωρήπανσης στις πόλεις. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω Εάν έχετε την πρόθεση να αναθεωρήσετε την Λευκή Βίβλο το επόμενο εξάμεινο, το προσεχής εξάμεινο και να εισαγάγετε αλλαγές ή τροποποιήσεις όσον αφορά την, ανάπτυξη, την αστική ανάπτυξη και τις μεταφορές. Και να πω ότι αναφέρομαι στα σχέδιά σας για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις πόλεις. Thank Σας ευχαριστώ. Η ευφυείς πόλης όπως σας είπα, θα είναι ένα πολύ ε, ενδιαφέρον στοιχείο. Θα, φυσικά θα συμμετέχω στην προσπάθεια στο μέλλον. Αν εγκριθεί η υποψηφιότητά μου, το ενδιαφέρον είναι ότι ε, συμπυκνώνονται διάφορες προσπάθειες σε ένα κοινό πρόγραμμα. Ε, η συμφόρηση είναι μεγάλη στα αστικά κέντρα, χρειάζεται καλύτερος σχεδιασμός για να αντιμετωπιστεί παραδείγματος χάρη το μεγάλο πρόβλημα της ρήπανσης όπως είπατε. Ο αστικός σχεδιασμός είναι παρόλα αυτά εθνικό ζήτημα. Βλέπουμε ότι επί τη βάση βελτίστων πρακτικών τα κράτη-μέλη εκδηλώνουν ένα ενδιαφέρον για έναν ευρωπαϊκό συντονισμό. Μου αρέσει το πρόγραμμα Ευφυής Πόλης διότι συλλέγονται οι διάφορες μετρήσεις Μαθαίνουμε έτσι πώς να αξιολογούμε καλύτερα και άρα και να αναλαμβάνουμε αποτελεσματικότερα μέτρα. Για την ηχορύπανση και την ρύπανση του αέρα, θα έλεγα ότι ε, μπλεκόμενοι φορείς όχι μόνο από τους τεχνικούς ε, τομείς αλλά και από ε, πολίτες θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι διότι πρέπει να αλλάξουμε και τις συνήθειές μας πέρα από το σχεδιασμό να ξέρουμε πού θα βάλουμε τα εργοστάσια, πού θα είναι τα γραφεία και οι επιχειρήσεις, πού θα είναι τα σπίτια δεν μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα το πρωί εξάλλου είδα ότι πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, ήμασταν σε μία λωρίδα όλοι, προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο αεροδρόμιο και τρεις λωρίδες παραδίπλα ήταν άδειε. Κάτι δεν πάει καλά με το σχεδιασμό. Θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλα όταν θέλουμε να παρεμβαίνουμε σε επίπεδο πόλης. Πρέπει να σας διακόψω, λέει ο πρόεδρος. Τρεις φορές σας έκανα νόημα, γι' αυτό πρέπει να το κάνω. Μην μου θυμώσετε λοιπόν. Επόμενη ερώτηση από την τύριο Δεκλούν για το ΕΛΚ. <laughs> Στην αρχική, στην αρχική σας δήλωση αναφερθήκατε στη βέλτιστη διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Περιφερειακά και τοπικά αεροδρόμια είναι ζωτικό σύνδεσμος με τον έξω κόσμο. Σημαντικά. Ε, προωθούν τον τουρισμό, τις επενδύσεις και είναι γραμμή ζωής για τις τοπικές κοινότητες. Χρησιμότατες υποδομές, πολύτιμες, πρέπει να προστατευτούν. Θα χαλαρωθούν οι κανόνες, θα χαλαρώσουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Πώς θα προστατεύσετε τα περιφερειακά αεροδρόμια και τι θα γίνεται με τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά, πώς θα καλύπτονται συγκοινωνιακά. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Σχετίζομαι με αυτό το θέμα, με απασχολεί αυτό το θέμα, με αρέσει, συμφωνώ μαζί σας και τα λιμάνια αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των ντόπιων περιοχών. Κυρίως από μακρισμένες περιοχές. Μου αρέσει να πετάω δεν θα είχα αυτή την πολιτισμική εμπειρία αν δεν χρησιμοποιούσα πτήσεις. Εάν δεν είχα πάει στις δυτικές ευρύδες αεροπορικά. Έχει πάρα πολύ, έχω πολύ ενδιαφέροντα αεροδρόμιο και στο Βάρα πήγα, στο σχετικό αεροδρόμιο και άμα αφησάει πολύ δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο. Είναι ζωτική σημασία για τις δυτικές ευρύδες, για τη Σκοτία, πολύ σημαντικό αεροδρόμιο. Πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα αεροδρόμια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και το εξής χρειάζεται οικονομική υποδομή. Θα μπορεί να συντηρείται από μόνο το τεροδρόμιο. Δεν μπορούν να, οι επιχορηγήσεις και η ενίσχυση να συνεχίζονται SAE. Είναι δύσκολο να μιλήσω για τις κρατικές ενισχύσεις, για τις ενισχύσεις γενικά. Δεν αποτελεί τμήμα των αρμοδιοτήτων μου. Όμως θα ήθελα να πω ότι είμαι πρόθυμη να συνομιλήσω με τους υπεύθυνους, να ακούσω την άποψή τους θα προσπαθήσω ε, να βρω νέα επιχειρηματικά μοντέλα που να συνδέονται πιο στενά με τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις έτσι αυτά τα σημαντικά αεροδρόμια να παραμείνουν ζωντανά. Είναι σημαντικά στις τοπικές κοινότητες της Σλοβενίας, το Πόρτο Ρος. Έχουμε ένα πολύ μικρό αεροδρόμιο, σημαντικότατο, για την άφηξη του κόσμου, των τουριστών από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη πρέπει να βρεθούν καλύτερες λύσεις. Αν μπορέσω, θα ήθελα και εγώ να μπορέσω να μεταβιβάσω τις εμπειρίες μου, τις σκέψεις μου για το νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Κύριος Πίτερ Βαντάν από το ECR έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Μιλήσατε για τις εσωτερικές πλωτές οδούς Υπάρχει ένα πρόβλημα. Με ένα τεχνικό πρόβλημα. Ακούτε τώρα. Ωραία. Ξαναρχίστε παρακαλώ. Καλησπέρα κυρία Μπούλτς. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μιλούσατε για την υποδομή που σχετίζεται με τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τη διασύνδεση ανάμεσα στις δυτικές και ανατολικές ε, πλωτές οδούς. Ε, στο Δούναβι, ανάμεσα στο Στρόπικινγκ, στο Βίλσαου ε, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Τι προτίθεστε να κάνετε ούτως ώστε να εξομαλυνθεί εκεί η μεταφορά στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Δεύτερον, μιλήσατε για την ενέργεια. Θα ήθελα να αναφερθώ στο EcoCombi. Κάποιοι μιλάνε για τα γιγαντία πλοία μεταφοράς κοντέινερ. Πολύ μεγάλα φορτηγά μεταφοράς κοντέινερς. Ε, εσείς τι έχετε να πείτε σε σχέση με τα EcoCombi. Απάντηση. Μιλάτε για αυτά τα τεράστια φορτηγά, σωστά. Ναι. Ας αρχίσω όμως με το Δούναβι. Ο Δούναβις ε, είναι πολύ σημαντικό τμήμα των σχεδίων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, πιστεύω ότι για τη διαβάθυνση του, ε, ε του Δούναβι θα μπορέσουμε να έχουμε τα ικανοποιητικά αποτελέσματα για να εξομαλυνθούν και οι μεταφορές από περιβαλλοντικής πλευράς είναι σημαντική η πρόκληση και θα πρέπει ε, να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα και να αντιμετωπίσουμε τις οικολογικές προκλήσεις. Πέραν αυτού δεν εμπλέκονται μόνο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο-τρεις χώρες ε, που συμμετέχουν ε, στο πρόγραμμα του Δούναβη θα χρειαστούν διμερείς και τριμερείς συζητήσεις για να επέλθει συμφωνία κυρίως για τη χρηματοδότηση. Έχει ήδη προγραμματιστεί ε, το θέμα του Δουναβή για τα διευρωπαϊκά για το βασικό κομμάτι των Ευρωπαϊκών αλλά δεν είναι μόνο δικό μας ζήτημα. Υπάρχουν και δύο-τρεις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση. Έχω ακούσει ότι είναι μεγάλη πρόκληση αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχα χρόνο για να διαμορφώσω άποψη. Εγώ θα έλεγα ότι θα παραμείνουμε ουδέτεροι και θα επιτρέψουμε, αλλά ποια είμαι εγώ για να επιτρέψω οτιδήποτε, θα, θα, νομίζω ότι κάποιοι, κάποιες χώρες θα ε, συνάψουν διμερείς συμφωνίες, αλλά δεν είναι πολύ ε, ευρωπαϊκή αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ. Λούση Άντερσεν από τους σοσιαλιστές. Μπορείτε να μας πείτε κυρία Μπούλς τι θα κάνετε τόσο ώστε όλοι οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και με ειδικές ανάγκες να έχουν ικανοποιητική πρόσβαση στα δίκτυα. Σας είπα, είπατε στην αρχή ότι εστιάζετε την προσοχή σας στους ανθρώπους. Τι εννοούσατε, θα ενημερώνονται οι άνθρωποι ε, για τα, τις, τις ε, μεταφορές και άλλα συναφή ζητήματα. Μίλησατε για τις αλλαγές. Ωραία. Ε, πολύ ωραία αυτά τα δίκτυα για τη διασύνδεση της Ευρώπης και η διάδρομη. Τι γίνεται όμως με τις εκατοντάδες χιλιάδες σταθμών και δικτύων όπου δεν υπάρχουν ασανσέρ και πρέπει να κουβαλάμε τις βαλίτσες μας ε, και υπάρχουν μόνο τα σκαλιά. Ε, όταν είναι ευρωπαϊκά τα κονδύλια, ασχολούμαστε με τα θέματα της μειωμένης κινητικότητας. Ο κύριος Βάντεν Κάμπ ε, δεν μας είπε τίποτα για αυτό το ζήτημα. Εσείς πώς θα μπορούσατε να επεκταθείτε. Απάντηση. Εάν θέλουμε να είμαστε στο πλευρό των επιβατών και να ακολουθήσουμε κοινωνικό προσανατολισμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα που εγείρεται. Ε, υπάρχουν ήδη ενισχύει οδηγίε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και στην πατρίδα μου μπορώ να σας πω ότι πριν από 10-15 χρόνια Κανείς ε, δεν είχε σκεφτεί να φτιάξει τις ειδικές ράμπες ε, στα λεωφορεία ε, για τους ΑΜΕΑ. Τώρα έχει ήδη συμβεί αυτό και σταδιακά θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες ε, οι ΑΜΕΑ. Ε, τώρα γίνεται νυχθημερών αυτό δεν νομίζω. Ασκώντας όμως διαρκή πίεση και φροντίζοντας να ακολουθήσουν όλο το καλό παράδειγμα κάνοντας ε, τους απαιτούμενους ε, ελέγχους και επιθεωρήσεις για να υπάρχει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία μπορούμε να το καταφέρουμε. Ε, αναφερθήκατε επίσης σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών. Πιστεύω με τα νέα προτινόμενα διαχειριστικά συστήματα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τα, ε, ε, ο κατακαιρματισμός των εθνικών συστημάτων διαχείρισης δεν επιτρέπει ε, καλύτερη ενημέρωση. Όμως με τα ενοποιημένα διαχειριστικά προγράμματα θα υπάρξει καλύτερη ενημέρωση όχι μόνο για τα εισιτήρια, για τις ε, συνθήκες, για τα δρομολόγια, Και αυτό καλύπτει φυσικά και ε, την ενημέρωση για τους ΑΜΕΑ που μπορούν ε, να ταξιδέψουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπιλμπάου Παραντίχα ε, από τους φιλελεύθερους τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε κύριε Προτινόμενη Επίτροπε, το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο προτάθηκε επειδή το τρίτο δεν είχε αποτελέσματα. Ε, τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να παρακάμψετε το μονοπόλιο των κρατών μελών και την αντίδρασή τους. Το Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει θέσεις πολιτικές για το σιδηροδρομικό πακέτο και ε, πολλές ε, εταιρείε και επιχειρήσεις θέλουν μείωση της γραφειοκρατίας και ασφάλεια. Εάν συνεχιστεί αυτή η στάση, εσείς πώς θα προχωρήσετε το θέμα της διαλειτουργικότητας, πώς θα το κάνετε αυτό χωρίς αυτή την πολιτική στήριξη και τι θα γίνει με την εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και τις επενδύσεις και πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ευβιωσιμότητας εάν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια. Επίσης, ο διαχωρισμός της διαχείρισης των υποδομών από τους παρόχους υπηρεσιών. Εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση και μακάρι να είχα πέντε λεπτά χρόνο για να απαντήσω. Όμως, να πω καταρχάς ότι θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά ως ένα ενιαίο πακέτο. Θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε το τεχνικό ε, επίπεδο, την τεχνική πτυχή και την πολιτική, θα την έλεγα εγώ πιο πολύ οικονομική πτυχή. Καταρχάς, το πρόγραμμα REFIT ενώνει πάρα πολλές διαφορετικές νομοθεσίες, πάρα πολλά έγγραφα και το πρόγραμμα REFIT θα απλοποιηθεί και θα γίνει πιο εύληπτο έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να καταλαβαίνει καλύτερα πότε δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του και ποια δικαιώματα πρέπει να ε, ποια δικαιώματα έχει και ποιες υποχρεώσεις έχει. Επίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το ανεξάρτητο δίκτυο διαχείρισης και διαλειτουργικότητας και εάν τα κρατημέλη δεν, ακόμα και αν τα κρατημέλη δεν το επιθυμούν, πρέπει να τα πιέσουμε να έχουν σαφείς και διάφανες ε, πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, υπολογίσουμε το κόστος ε, μιας υπηρεσίας. Διαφορετικά δεν μπορούμε. Ήμουν για πάρα πολλά χρόνια διευθύντρια μιας μικρής εταιρείας και επίσης διευθύντρια των τηλεπικοινωνιών στην Σλοβενία. Και πραγματικά μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι αν δεν ξέρεις το πραγματικό κόστος μιας υπηρεσία που παρέχει, δεν μπορεί να κάνεις ε, καμία σωστή διαχείριση και δεν μπορείς να λάβεις καμία σωστή απόφαση για τη διαχείριση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το πακέτο και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αν και να πω ότι το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει θετικά στην πρώτη φάση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μην το διαχωρίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά ενωμένο, διότι θέλουμε να απελευθερώσουμε την αγορά και να την κάνουμε πιο προσιτή. Ο επόμενος ο, ομιλητής είναι Λούις Πασκουάλ από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το πρόβλημα που έχει προκύψει. Έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες για μεταφορές επιβατών και για ταξί στις ε, πόλεις και σίγουρα απαιτούνται κάποιες άδειες και κάποια ασφάλιση για να γίνει αυτό, κάποιες ε, φορολογικές ε, δηλώσεις όταν αυτές οι εταιρείες ταξί, οι ιδιωτικές εταιρείες ταξί δεν ε, πληρούν τις ε, προϋποθέσεις, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, ποια μέτρα ε, θέλετε εσείς να λάβετε στον τομέα αυτό και αν υπάρχει κάποια συντονισμένη δράση από πλευράς ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να τη στηρίζουν και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αποτρέψουν τον αθέμητο ανταγωνισμό και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Έπειτα για τον έμπολα. Η επιδημία αυτή του έμπολα έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες. Και υπάρχει και μια πρόσφατη σύνοδο κορυφής η οποία αποφάσισε να βελτιωθεί η εναέρια κυκλοφορία. Εσείς όμως ανεξάρτητα από τα κράτη-μέλη τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου στα αεροδρόμια για να καταπολεμηθεί ο έμπολα. Ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις σας. Η πρώτη ερώτηση που θέσατε υποστηρίζω αυτά που ήδη προτείνατε στην ερώτησή σας. Θα πρέπει να έχουμε σαφή διοργάνωση. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες όταν πήγα στις Βρυξέλλες έπαιρνα ένα ταξί που αναφερθήκα στα ταξί και υπάρχει νέα απέτηση θα πρέπει να έχουν οι ταξιτζίδες αριθμούς που φαίνονται καθαρά θα πρέπει να καταβάλουν τέλη μηνιαίως για τη λειτουργία του ταξί. Στην αρχή η οδηγή των ταξί παραπονιότανε. Τον ρώτησα μου στον οδηγό συγκεκριμένο συγκεκριμένου, σας αρέσει. Τον ρώτησα, μου λέει ναι, το μόνο το οποίο παραπονιόμαι, παραπονέθηκα στην αρχή γιατί είπα να πληρώσω 200 ευρώ για την άδεια και και τώρα η άδεια έχει γίνει 50. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όλα τα άλλα είναι δίκαια, είπε ο οδηγός. Ποια είναι η απάντησή μου είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη. Είναι τοπικό θέμα. Μπορούμε να βοηθήσουμε όμως, να στηρίξουμε το μέτρο, να το προωθήσουμε και αν βρούμε κάποια στοιχεία που είναι κοινά για όλη την Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, οπωσδήποτε πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις, ε, όλα τα μέτρα που καταπολεμούν τον τον ανταγωνισμό για την έμπολα δεν πρέπει να κρίσουν οι διάφορες εγκαταστάσεις οπότε δεν μπορούμε να ενεργοποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Χρειάζεται όμως μια ευρωπαϊκή τοποθέτηση γι' αυτό. Είναι Σαγιάζα Σέντερ για τους σοσιαλιστές. επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, πρώτα απ' όλα εκφράζω ικανοποίηση διότι έχετε βολή, έχετε μπει σε μαραθώνη. σας θαυμάζω για την ετοιμασία που κάνατε για το μαραθώνι αυτόν τον οποίο ζείτε. Λοιπόν, για τις υποδομές ήμουν εισηγήτρια ε, για τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν τα δίκτυα για όλες τις ανάγκες το, για τις βιώσιμες μεταφορές στην Ευρώπη. Φαίνεται μικρό το ποσό αυτό και η πρόκληση είναι να χρησιμοποιηθούν πολύ σωστά οι διαθέσιμοι πόροι. Είπατε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα διάφορα μέσα. Υπάρχουν εμπόδια όμως και κυρίως πρόκειται για συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα και τα κράτη-μέλη τα περισσότερα έχουν πρόβλημα όσον αφορά το δημόσιο χρέος και δεν έχουν χρήματα για τη συγχρηματοδότηση. Λοιπόν, χρειάζεται μια κάποια ευελιξία και θα ήθελα να γνωρίζω αν εσείς με τον Κατάνιο και τον Μοσκοβιτσί θα μπορέσετε να βοηθήσετε τις χώρες ούτως ώστε οι επενδύσει τις ε, υποδομές να μην αυξήσουν σημαντικά το δημόσιο χρέος. Άλλο εμπόδιο είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε διμερές επίπεδο. Είμαι Ισπανίδα και εμείς θα θέλαμε να, να περάσουμε τα πυρηναία, να διασχίσουμε τα πυρηναία και οι Γάλλοι δεν το θέλουν ε, υπάρχει ένας υπέροχος κανονισμός της Ευρώπης και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα διέξοδο. Τι θα κάνει η Βρυξέλλες, τι θα κάνει η Βρυξέλλες το θέμα. Κοινωνικό πακέτο, αναφερθήκατε στη Λευκή Βίβλο, είναι μακροσκελή έγγραφα οι Λευκές Βίβλοι, περίπλοκα χρήμα, ε, έγγραφα. Είναι αρχές που αναφέρονται. Εμεί χρειαζόμαστε δράσεις και όχι απλώς αρχές που αναφέρονται σε κάποια έγγραφα. Δεν υπάρχουν και κεφάλαια. Λοιπόν, και οδηγεί τον ε, φορτηγών ε, γυράσκουν. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό πακέτο για τις μεταφορές. Θα το διαπραγματευτείτε αυτό. Είχατε τρία λεπτά. Χρησιμοποίησατε τα δύο. Σας μένει ένα. Παρακαλώ απαντήστε. Καλώς, πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις υποδομές που αναφερατε, όπως προανέφερα, ναι, θα χρειαστούμε καινοτόμου οικονομικούς μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση. Δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας να χρηματοδοτήσουμε τα πάντα. Είναι γεγονός. Πώς θα τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολο να πω τώρα. Ε, ίσως θα ήταν άδικο να κάνω κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι αν εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι από τις σοβαρότερες συζητήσεις που πρέπει να διεξαχθούν θα πρέπει να ξεκινήσουμε σοβαρό προβληματισμό, να, καλές, να προσελκύσουμε και επενδυτέ στον ιδιωτικό τομέα. Άκουσα χτε διάβασα στο Financial Times ότι ήδη γίνονται προσπάθειε να συμμετάσχουν τα συνταξιωτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία. Άρα υπάρχουν πάρα πολλέ ευκαιρίε. Είναι σοβαρή πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Μπάχ, το λέω από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αποψήφια Επίτροπε. Με εντυπωσίασαν όλα όσα είπατε. Δύο όμως ε, πάνω απ' όλα. Καταρχάς ε, οι άνθρωποι και το ε, ενδιαφέρον που δίνετε κυρίως στους ανθρώπους και το ενδιαφέρον για το διάλογο που έχετε. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών, ακριβώς όπως και η ερώτηση της κυρίας Άντερσον. Θα, εσείς σε ενδεχόμενη επανεπεξεργασία της σχετικής ε, νομοθεσίας θα θέσετε τον επιβάτη στο προσκήνιο και έπειτα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορες στις ε, απόψεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και επίσης ότι υπάρχει έλλειψη νομικής διαφάνειας και γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αναγκασμένο να κάνει τη δική μας δουλειά. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να βγάλετε από το αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε η νομοθετική αρμοδιότητα να επιστρέψει ξανά στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο από τη δική σας πλευρά ως υποψήφια επίτροπος. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Καταρχάς, δικαιώματα των επιβατών και αυτό είναι ένα τεράστιο πίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ετοιμάσει ένα πραγματικά εξαιρετικό πακέτο για τα δικαιώματα των επιβατών. Ωστόσο, παρατηρώ ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προτιμούν να κυρώσουν μία πτήση παρά να ακολουθήσουν συστάσεις ή κανόνες που εφαρμόζονται. Εμείς θέλουμε να το αποτρέψουμε αυτό. Δεν έχω τώρα κάποια απάντηση και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας και αυτό διότι δεν γνωρίζω ακριβώς πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι πολύ ψηλά στις δικές μου προτεραιότητες. Είμαι και εγώ επιβάτης και ξέρω από πρώτο χέρι ε, τι συμβαίνει και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Πιστεύω λοιπόν σε έναν επικοδομητικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και να μην μείνουμε μόνο στα δικά μας σύνορα αλλά να ε, επεκτείνουμε τα δικαιώματα των επιβατών και εκτός ευρωπαϊκών σύνορων. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω ε, την ερώτηση σχετικά με το Γιβραλτάρ που είχατε πει. Πιστεύω πως το ερώτημα είναι πολιτικό και δεν θα έπρεπε να καθυστερεί αυτό τις αποφάσεις θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθούμε στις, στα έργα και να δούμε όταν θα επιληθεί το ζήτημα τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαλτέζ έχει το λόγο. Κυρία Επίτροπε, ήμουν προλίγου στη Τζένοβα που έχει ζήσει τη δραματική κατάσταση των πλημμυρών. Είναι δύσκολο να πώ στου πολίτε τη πόλη εξακολουθεί να εξοδεύει δισεκατομμύρια στα έργα Ευρώπη και δεν καταφέρνει να βρει λίγα εκατομμύρια να αποφευθεί η τραγωδία όπω αυτή που συνέβη στη Τζένοβα. Σήμερα έχει ένα σύστημα κυβέρνηση για τα ύδατα που είναι λιγότερο αποτελεσματικό από αυτό που είχε το 15ο αιώνο. Λοιπόν, λόγω περικοπών. Θα επανεξετάσετε λοιπόν τι αποφάσει του 2013 και να καταργηθούν κάποια από τα άχρηστα έργα που κινδυνεύουν να επιδεινώσουν ε, την υδρογεολογική σταθερότητα σε διάφορε περιφερειε της Ευρώπης. Ήδη όπω δείχνουν και πλημμύρε στην Ιταλία ε, και πριν στην Βρετανία, στη Γερμανία και στη Τσεχική Δημοκρατία. Υπάρχουν προβλήματα. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν προτίθεστε να αναλύσετε πριν ξεκινήσουν κάποιοι διαγωνισμοί από τα μεγάλα έργα που υπάρχουν όπως το Ρήνο Λιόν. Η γραμμή αυτή κοστίζει, είναι το πιο δαπανηρό έργο. 150 ε, εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο κοστίζει ε, και μήπως θα πρέπει να γίνουν νέες μελέτες για το συγκεκριμένο έργο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι πλημμύρες είναι πολύ ατυχή συμβάντα και η χώρα μου έχει πληγεί σοβαρά από αυτές. Αλλά τι βλέπουμε, ότι δεν είναι ένα πρόβλημα της χώρες όπου εμφανίζονται οι πλημμύρες, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αφορά το όλο υδάτινο σύστημα, διότι κάπου το νερό θέλει να περάσει. Διότι σωρεύεται σε ποσότητες στη διαδρομή που ακολουθεί. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι στο ΣΕΦ ήδη ε, έχουμε θέσει προτεραιότητες, έχουν καλυφθεί κάποιες προτεραιότητες για να αποφευχθούν στο, μέρος, στο μέλλον οι πλημμύρες. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ευπρόσδεκτες περαιτέρω συζητήσεις για τις πλημμύρες δεν μπορώ να δεσμευτώ πέρα από αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Όλα αυτά αφορούν τη ζωή. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε με κάτι που εγκρίθηκε πριν από χρόνια, όταν α, μας προβάλλει προκλήσει ζωή. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Καλωσορίζω περαιτέρω συζητήσεις. Ελπίζω ότι ό,τι έχει εγκριθεί να επανεξεταστεί, να προωθηθεί για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Αυτή δεν ήταν η μόνη ερώτηση που είχατε θέσει από την πλευρά σας, έτσι δεν είναι. Επόμενος ο Ντάφορ Σκέρλετς από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Μπούλτς, η δημόσια υγεία και η πολιτική μεταφορών συνδέονται στενά. Παραδείγματος χάρη, η η χορύπανση οδηγεί σε διατάραξη των οικοσυστημάτων. Επίσης, ε, δεν υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση πώς επηρεάζει η πολιτική μεταφορών ε, την ε, ποιότητα ζωής, ε, τις κλιματικές αλλαγές, τις, την ανθρώπινη υγεία, οι καρδιακιακές επαθήσεις, παραδείγματος χάρη, συνδέονται με τις μεταφορές, επιζήμιες επιπτώσεις των εναερίων μεταφορών, με πάρα πολλούς τρόπους πλήττεται η ανθρώπινη υγεία από τα διάφορα είδη μεταφορών. Ποια μέτρα θα αναλάβετε το ώστε τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας να ενσωματωθούν στον τομέα των μεταφορών. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πιστεύω ότι στη σύγχρονη κοινωνία συνειδητοποιούμε όλη αυτή την πρόκληση και έχουν πολλαπλασιαστεί τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής πέρα από την ανθρώπινη υγεία. Δεν θα τα επαναλάβω αυτό που μας είπατε στην ερώτησή σας. Με ρωτήσατε τι θα κάνω. Ναι, ποτέ δεν αρκούν οι προσπάθειές μας. Δεν μπορεί να αρκέσουν οι προσπάθειες σε καμία περίπτωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Ε, ξέρω πόσο επιζήμια είναι η χορύπανση ε, στον τομέα των συνδρομικών μεταφορών και οδικών μεταφορών υπάρχουν νέα συστήματα πέδησης παραδείγματο χάρη που μειώνουν την ηχορύπανση. Δεν είναι η τέλεια λύση, αλλά είναι μία πρόοδος. Οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν. Θα έχουμε πιο σιωπηρά μηχανήματα, διαφορετικούς κινητήρες, αν χρησιμοποιούμε άλλες ενεργειακές πηγές. Και αυτό θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων τα θύματα της σύγχρονης ζωής, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Πολύ καλή ερώτηση. Μέσα από τον κοινωνικό διάλογο μπορούμε να βρούμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Αστικός πολεδομικός ε, σχεδιασμός δεν είναι μόνο ε, ε, δική μου αρμοδιότητα, δεν σχετίζεται μόνο με το δικό μου χαρτοφυλάκι των μεταφορών θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις που περιγράψονται. Σας ευχαριστούμε Γιώργ Μάιερ, ε, μη γραμμένος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπούλκ, εδώ μπροστά σας είμαι. Καλώ ήλθατε λοιπόν. Ω Αυστριακό είμαι και γείτονά σα και θα ήθελα λοιπόν να σα καλωσορίσω και να σα ε, απευθύνω μια ερώτηση ω άμεσο γείτονά σα. Είμαι από τον Κράτ και τον Κράτ δεν απέχει και πολύ από τη Σλοβενία. Και να σας ερωτήσω λοιπόν το εξής. Χαίρομαι πολύ με το ότι παραδέχεστε τις αδυναμίες σας, ότι λέτε πως δεν γνωρίζετε κάτι. Όσον αφορά τώρα τον ε, διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής, ε, ίσως ε, θα έχετε ενημερωθεί ότι από την, ε, από την διεύρυνση του 2004 η Αυστρία έχει γίνει χώρα διέλευσης. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφώνηση και ε, αυτός ο άξονας έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Εσείς τι ε, σχέδια έχετε, εάν είναι φυσικά οικονομικά εφικτό, έτσι ώστε να ελαφρύνετε την συμφόρηση που παρατηρείτε εσεί στην περιοχή. Είναι κάτι που αφορά την Αυστρία, αλλά όχι μόνο την Αυστρία. Και ε, κάνω την ερώτηση σε εσά, ε, διότι είστε, πιστεύω, και η πιο αρμοδία να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για τις προτεραιότητες και όλους τους διαδρόμους έχουν εγκριθεί τα σχέδια από το CEF. Ε, ό,τι είχε εγκριθεί στα πλαίσια των διευρωπαϊκών θα το υποστηρίξω, θα το προωθήσω. Εξυπακούεται. Εγώ γνωρίζω την περίπτωση της Σλοβενίας. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για να ακολουθηθούν αυτοί, αυτές οι προδιαγεγραμμένες ε, διαδρομές. Ε, η Σλοβενία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, το κάνει για το πακέτο 1, αφήστε το πακέτο 2 και 3. Είναι μεγάλε οι προκλήσει ακόμη και για τα προηγούμενα πακέτα. Ελπίζω να μην προκύψει και πακέτο 5. Ελπίζω να παραμείνουμε στα 3 και 4 προς το παρόν. Τι μπορώ να σας πω. Θα ακολουθήσω στο μέτρο δυνατό τις προτεραιότητες του CEF και οι χώρες που είναι στους βασικούς διαδρόμους θα φροντίσω να συμμορφωθούν με τα υπεσχημένα, με τα ε, στοιχεία των προηγουμένων ε, πακέτων. Ε, για το διάδρομο των Βαλκανίων θα δούμε ποια επιτυχία θα έχει και με τη δική σας βοήθεια ελπίζω να αυξηθεί η πίεση προς τις χώρες ε, για να συμμορφωθούν με τις ε, προηγούμενους, ε, από τα προηγούμενα πακέτα. Καλόν που φορά από τους σοσιαλιστές οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί στα πλαίσια τη συνολική προσπάθεια των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των δαπάνων πρέπει να μειώσουν κατά 5% τα έξοδά του. Ο, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδροδρόμων όμω θα, πρέπει ε, να έχει αυξημένε αρμοδιότητε. Ε, με περιορισμένα μέσα και με περιορισμένο προσωπικό θα μπορέσει να αντεπεξέλθει. Ο Μάρκο Εύκοβιτ στην ακρόαση τη 30 Σεπτεμβρίου ανέλαβε δέσμευση να, ε, για την αύξηση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ιδροδρόμων κυρίω με απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμών. Θα τηρήσετε αυτή τη δέσμευση. Αυτό σημαίνει αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ή ανακατανομή των ε, κονδυλίων που έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, ε, ερώτησή σας. Θα, το αφεντικό μου θα είναι ο κύριος Εύκοβιτς, εκείνος θα συντονίζει, οπότε έχω κάθε συμφέρον να ε, ακολουθήσω αυτά που προτείνει. Για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, υπάρχουν δύο όψεις σε αυτή την ερώτηση. Και θα φτάσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Το πρώτο γενικότερο θέμα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν γενικότερα οι οργανισμοί. Έχει συμφωνηθεί και έχουμε κάποια καλά παραδείγματα εξωτερικής ανάθεσης των υπηρεσιών των οργανισμών. Δηλαδή θα πρέπει να ε, επιδιώκουν να έχουν υπηρεσίες στις οποίες θα μπορούν να συγχρηματοδοτούν Αυτό όμως δεν απαντά στην ερώτησή σας. Τι γίνεται όταν αυξάνονται οι αρμοδιότητες των οργανισμών και μειώνονται τα μέσα. Αυτό ισχύει για όλες τις διοικήσεις, ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και στη Σλοβενία το ίδιο σημαίνει. Πρέπει να περικόψουμε το κόστος της διοίκησης για μια σύγχρονη οικονομία είναι υπερβολικό το κόστος και δεν μπορεί πλέον να απορροφηθεί. Ωραία. Απ' την άλλη όταν ε, είναι αυξημένες και νομιμοποιούνται οι αυξημένες αρμοδιότητες θα αγωνιστούμε για τα απαιτούμενα κονδύλια, τα κονδύλια που απαιτούνται για να επιτελέσουν οι οργανισμοί το έργο που τους ανατίθεται. Κυρία Σμιτ, ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό για να μπορέσει να υπάρξει ενιαίος οικονομικός χώρος. είναι γνωστές οι άποψή σας για αυτό το, θέμα και δεν είμαι η μόνη που τον, τις καλωσορίζω άλλωστε. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερα από λόγια και περισσότερα ε, πράγματα από προσπάθειες και ε, ωραίες διατυπώσεις. Υπάρχουν 23 διαφορετικά συστήματα για τα διόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από τις γερμανικές συζητήσεις για τα διόδια έχει ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας που είναι δύσκολο να κλείσει. Τα διόδια σίγουρα μπορούν να επιφέρουν ε, προστιθέμενη αξία και να κλείσουν ορισμένες ε, τρύπες ε, του προϋπολογισμού. Όμως για να γίνει αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί φόροι. Ε, εάν όντως γίνουν επενδύσεις στις υποδομές δεν θα είχαμε προβλήματα και δεν θα χρειαζόταν τρομακτική βελτίωση για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Εσείς τονίσατε την δική σας εμπειρία από τις μεταφορές και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την πολιτική μεταφορών. Πώς λοιπόν ε, σκοπεύετε να ενώσετε αυτά τα 23 διαφορετικά συστήματα διοδίων και να τα ενώσετε σε ένα ενιαίο σύστημα διοδίων το οποίο σκοπό θα έχει να δώσει έσοδα για ε, επενδύσεις στις υποδομές και να ε, αυξήσει την ταχύτητα της κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκές οδούς. Ξανά θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη στην απάντησή μου. Καταρχάς ήδη έχουμε συμφωνήσει και στηρίζω αυτή τη θέση. Συμφωνήσαμε ότι θα εφαρμόσουμε τον κανόνα σύμφωνα τον οποίο ο χρήστης πληρώνει και ο ρηπαίνων πληρώνει. Τι σημαίνει αυτό για τα συστήματα διοδίων. Τα συστήματα των διοδίων είναι θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς την τιμή αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε ότι να βασίζεται η τιμή επί του κόστους. Και θα επιμείνω από αυτού. Τιμολόγηση με βάση το κόστος είναι πολύ καλή λύση. Δεν μπορούμε όμως να συγκρίνουμε τις τιμές που προβλέπονται στις διάφορες χώρες. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Μακροπρόθεσμο όραμά μου ποιο είναι. Αν έχουμε ενοποιημένο σύστημα που και τα όλα έχουν απεμπλακεί και έχουμε σαφή λογιστικά στοιχεία και μπορούμε να δούμε την τιμολόγηση, τις τιμές, τη συμπερίληψη εξωτερικών τιμών κλπ. θα ήταν καλά, αλλά είναι μακροπρόθεσμος στόχος. Θα ήθελα να κινηθούμε προς τα εκεί, διότι έτσι οι μεταφορές θα γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν είναι κάτι προβλέψιμο αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πολεμούσα τώρα για την τιμολόγηση βάση κόστους κάθε χώρα πραγματικά να απομακρυνθεί από διακριτικά στοιχεία που εφαρμόζονται. Ρόμπερτ Ζήλε, Ευχαριστώ. Πριν από κάποια χρόνια συζητούσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ευρωπαϊκά δίκτυα και το μέσο για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Και δεχτήκαμε τον, τον, τον κύριο Γιακούνη, επικεφαλής του ρωσικού μεταφορέα που ήθελε να γεφυρώσει την Ευρώπη με την Ασία και συνεργασία με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Εκεί συζητήθηκε και ένα πρόγραμμα για επέκταση των γραμμών των 50 μιλιμέτρων για από τα Ουκρανικά σύνορα προς Σλοβακία κλπ. Δηλαδή οι ράγες με μεγαλύτερη, μεγαλύτερο εύρος και κάποιες εταιρείε των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έκαναν κάποιες μελέτες. Ποια είναι η άποψή σας για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επεκταθούν ε, τα 15 με 20 αυτές οι ράγες, οι πιο φαρδιές στο δίκτυο της Ευρώπης αισθάνομαι, απάντηση ότι είναι καυτό θέμα αυτό θα είμαι πολύ ρεαλιστική δεν θα σας αρέσει η απάντηση αλλά δεν μπορώ να σας δώσω καλύτερη προτεραιότητες έχουν καθοριστεί στο μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπης, το CEF. Και θέλω να παραμείνουν σε αυτά τα πλαίσια. Όμως, αν η ευρωπαϊκή ραχοκοκαλιά θέλουμε να πετύχει, θα πρέπει να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο. Θα πρέπει να βρούμε νέες λύσεις για χρηματοδότηση, για συνεργασία, μέσω διμερών ε, συμφωνιών, ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων χωρών, ούτως ώστε το δίκτυό μας να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο σύστημα σιδηροδρομικό ή οδικό. Ήμουν πολύ ενθουσιώδης. Πριν από δύο μέρες το πρωινό διάβασα ένα άρθρο για διασύνδεση Κίνας και Ευρώπης, σιδηροδρομικής. Και πόσο υποφελές οικονομικά είναι αυτό. Είναι προγράμματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι 25% πιο ακριβά να ταξιδέψει κανείς σιδηροδρομικά από ό,τι με πλοίο. Αλλά χρειάζεται μόνο ένα μήνα εν συγκρίση με δύο μήνες με τον άλλο τρόπο. Άρα ε, είναι πολύ ελκυστικό η μεταφορά των προϊόντων. Οι σιδηρόδρομοι εδώ αρχίζουν να ανταγωνίζονται με άλλους τρόπους μεταφορών για τη μεταφορά αγαθών. Και σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει ο ανταγωνισμός. Πρέπει να το ξαναεξετάσουμε. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις, να βρούμε τρόπους για συγχρηματοδότηση των μέτρων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της. Γιάννης Νίλσον, επόμενος για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα ζήτημα που αναφέρθηκε ήδη, αλλά νομίζω ότι μπορεί να διασαφανιστεί. Ε, για τις παγκόσμιες μεταφορές ε, χρειαζόμαστε κανόνες για ανταγωνισμό επί τη βάση της ποιότητας, όχι με χαμηλούς μισθούς και κακές συνθήκες εργασίας. Οι φυστάμενοι κανόνες που κατοχυρούν τα κοινωνικά δικαιώματα, οι συλλογικέ κλαδικές συμβάσεις ε, δεν επαρκούν. Παραδείγματο χάρη ο χρόνος ε, ανάπαυσης. Ε, τι γίνεται με την εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών, πώς θα καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, είναι για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ποιες πρωτοβουλίες πρωτοβουλίε θα αναλάβει ε, ούτω ώστε να ε, την παράνομη ε, διακίνηση, το καμποτάζ, ε, τις παρατυπίες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Very serious uh, challenge. Πολύ σοβαρές οι προκλήσεις αυτές. Το παραδέχομαι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρία ερωτήματα για τον ανταγωνισμό πρώτα απ' όλα. Πάντοτε θα αγωνίζεται για θεμητούς όρους ανταγωνισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ε, τα κράτη-μέλη στο επίπεδο τους μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συνεργάζονται. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Θα το ενθαρρύνουμε, θα, θα το προωθήσουμε. Αναφέρθηκατε στο dumping. Πώς μπορούμε εμείς να εμποδίσουμε αυτές τις ε, ε, εταιρείες γραμματοκιβωτίου, τις εταιρείες βιτρίνα. Δεν μπορούμε όμως με κατάλληλη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, με αποκάλυψη των ε, παράτιμων αυτών επιχειρήσεων, κάνουμε ήδη ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το θέμα του καμποτάζ συνδέεται με την πράσινη ατζέντα. Με αυτά που προσπαθούμε, τα στοιχεία προσπαθούμε να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα φορτηγά πρέπει να είναι γεμάτα, φορτωμένα. Δεν έχει κανένα νόημα να ε, γυρνάνε άδεια. Βέβαια υπάρχει ο κανόνας των τριών γύρων πρωτού γυρίσουν στην χώρα προέλευσης. Θα πρέπει να δούμε αν αυτός ο κανόνας ε, συμβαδίζει με την ανταγωνιστικότητα που θέλουμε να επιτύχουμε χάρη στο πράσινο θεματολόγια. Πολύ μεγάλες αυτές οι προκλήσεις και διαρκώς θα μας ε, απασχολούν. Ευχαριστούμε. Άντρου Ντέλη από το ΕΛΚΑ. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μπούλτς, στην εισαγωγική σας παρουσίαση τονίσατε πόσο σημαντική είναι η διάδρομη των διευρωπαϊκών δικτύων για σας. Αυτή η διάδρομη είναι ε, σημαντική διεύλη επικοινωνία ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Έχουμε την στρατηγική του Δούναβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στόχο έχει να βελτιώσει την κινητικότητα στις ε, εσωτερικές πλωτούς, πλωτές οδούς. Όμως, δεν σταματάνε αυτές ε, στα εξωτερικά μας σύνορα, δηλαδή Ουκρανία, Σερβία, εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια. Πώς λοιπόν οι παραδουνάβιες χώρες αυτές θα μπορέσουν να βρούνε την κατάλληλη χρηματοδότηση για να επιτύχει η προσπάθειά μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, στο, στη Σλοβενία τι γίνεται με τους ποταμούς Λάβα και Ντράβα. Πρόκειται για άλλη διάσταση της, ε, των μεταφορών σε εσωτερικές πλωτούς όδους. Τι κάνει η Σλοβενία. Απάντηση. Σωστά το είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διάδρομη των διευρωπαϊκών δικτύων και εσωτερικές πλωτές οδοί είναι ένα απόσπαστο κομμάτι μεγαλύτερων δικτύων ε, που ε, συναποτελούνται από σιδηροδρόμους, οδικούς άξονες. Θα πρέπει με συστημικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προγράμματα. Μιλήσατε για τις παραδουνάβιες χώρες. Βεβαίως, μπλέκονται πάρα πολλές χώρες και όπως έλεγα, αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να προσκαλέσω όλους τους ενδιαφερομένους για να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης. Δεν μπορεί να τα Χρηματοπαϊκή Ένωση στο Ταμείο Συνοχής και στο CEF υπάρχουν κάποια διαθέσιμα κονδύλια για να βελτιώσουν τα κράτη-μέλη τις μεταφορές στις δικές τους εσωτερικές πλωτές οδούς, αλλά δεν επαρκούν αυτά τα κονδύλια πρέπει. Ε, σε χώρες που αναφέρατε και εσείς, στη Σερβία, στη Μολδαβία και Ουκρανία, μέχρι που φτάνουμε και στην, στον έξινο πόντο, να δούμε πώς θα ε, συνδυαστεί ε, συνδυαστούν οι ξένες άμεσες επενδύσεις με νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνεργασία χρειάζεται για να τα καταφέρουμε και το συνολικότερο δίκτυο μεταφορών ε, της Ευρώπης ε, βασίζεται και στους εταιρικές πρωτοσόδους. Ο Ντομινίκ Ρίκε, και πίσω σας, ε, Επιτρόπε. Πίσω σας είμαι, Επιτρόπε. Η οδηγία για τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους είναι πάρα πολύ σημαντική διότι συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όμως για πολλές ε, αρνητικές παράπλευρες επιπτώσεις. Ε, είναι ιδιάζνο με τομέας των μεταφορών διότι μετατοπίζονται, δεν αποσπονται οι εργαζόμενοι και προέκυψε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Στον τομέα των μεταφορών προτίθεστε να προωθήσετε αναθεώρηση, αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τους αποσπασμένους εργαζομένους γιατί οι αναθεωρήσεις που έγιναν δεν έλυσαν το πρόβλημα. Δεύτερον, σε σχέση με την απάντηση που μας δώσατε προ ολίγου, θέλετε να απελευθερώσετε δηλαδή παντελώς το δικό καμποτάζ αυτό μας λέτε. Τρίτον, για ε, ε υπάρχει περίπτωση ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ιδιαίτερα για το θέμα των ειδικών μεταφορών να συσταθεί ή να υπάρξει μια ε, διάσταση για τις οδικές μεταφορές σε έναν υφιστάμενο ευρωπαϊκό οργανισμό. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ε, ναι, ε, θα πρέπει να αναλυθεί το ζήτημα και θα το υποστηρίξω. Θα υποστηρίξω αυτή την ιδέα που υποδείξατε στην ερώτησή σας. Θα ήθελα να μάθω ποιε είναι οι παράπλευρες επιπτώσεις τη οδηγία για τους αποσπασμένου εργαζομένους ε, για να λυθεί το πρόβλημα κάποια στιγμή στο μέλλον. Για το οδικό καμποτάζ πιστεύω ότι υπάρχει στο τραπέζι μια συμφωνία. Εγώ αυτό που είχα κατά νου είναι να δούμε, να διαπιστώσουμε αν χρειάζεται διαρκής επανεξιολόγηση των κανόνων της νομοθεσίας. Αν κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί, τότε θα υποστηρίξω μια τέτοια ιδέα για έναν οργανισμό τώρα για τις οδικές μεταφορές. Όταν μιλάμε για τις ε, προκλήσεις και τις ευκαιρίες των οδικών μεταφορών, συνειδητοποιούμε ότι μόνο για αυτό τον τομέα δεν υπάρχει ειδικό οργανισμός. δεν ε, θα ήθελα να ε, σπεύσω, να συμφωνήσω με αυτή την, την καταφάνως καλή ιδέα. Ίσως θα ήταν ε, καλύτερο να ένα τμήμα ενός φυστάμενου οργανισμού να ασχοληθεί με τις οδικές μεταφορές. Sí, Καλημέρα, λέει ο μιλητή. Συγχαρητήρια και καλή τύχη, όπω λέμε στην Ιταλία. Η ερώτησή μου διαθρώνεται επί δύο ζητημάτων πολύ επικέρων και συντόμων. Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Συνδρομικής Κυκλοφορίας και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία της Διδροδρόμους. Για το πρώτο θέμα έχουμε αυτό το σύστημα που γεννάται με σκοπό να ενοποιήσει το ευρωπαϊκό σύστημα να εφαρμοστεί η ενωτική πτυχή. Αναφέρθηκε αυτό σε διάφορες ερωτήσεις, θετικές συνέπειες της διαλειτουργικότητας. Πάνω σε αυτό έχουμε τεχνικό ερώτημα. Τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αποφασιστούν, να καθοριστούν, να εφαρμοστούν. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν αφορά τη συνεισφορά που μπορείτε να κάνετε ούτως ώστε να υπάρξει σταθεροποίηση και αυτή η εξέλιξη. Μετά όσον αφορά την Ευρωπαϊκό Οργανισμό, Ευρωπαϊκό Οργανισμό, σας ρωτώ απευθείας, μπορείτε να συμβάλλετε στη αδειοδότηση και για τις σιδηροτροχές, και τον εξοπλισμό που τοποθετείτε στα τρένα να ανατεθεί στον οργανισμό. Και μια πατριωτική ερώτηση που αφορά την Ιταλία. Το σύστημα εσωτερικής ναυσοπλοείας αφορά και το μέλλον της Ιταλίας και το πιο σημαντικό ποτάμο, τον Πάδο. Λοιπόν, σας ρωτώ, θα μπορείτε να μας βοηθήσετε να ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά εμπόδια που μας εμπόδισαν ούτως ώστε να χρησιμοποιείται και στην Ιταλία η εσωτερική ναυσιπλοεία και να μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας η ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοείας στην Ιταλία. Μπορείτε να βοηθήσετε. Okay. Απάντηση. Καταρχάς σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Θα δούμε μέχρι πού μπορώ να προχωρήσω με τις απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα ο οργανισμός των σιδηροδρόμων. Ο οργανισμός των σιδηροδρόμων ήδη έχει παίξει απίστευτο ρόλο και έτσι όπως κινούμεθα που θέλουμε να ενοποιήσουμε το σιδηροδρομικό σύστημα θα γίνει πιο σημαντικός οργανισμός. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερες προδιαγραφές, πρότυπα, για τον εξοπλισμό, αλλά όχι μόνο για θέματα διασυνοριακής διασυνδημότητας, αλλά μεταξύ τοπικών ε, συστημάτων στιδρομικών και της βασικής ράχοκοκαλιάς. Εκεί μπορεί να παίξει ρόλο ο οργανισμός. Απ' την άλλη, έχουμε... Ε, κάπου έχασα τη σκέψη μου. Το είχα στο μυαλό μου, εδώ το είχα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα... Α, ναι, ο οργανισμός βοηθά τον καθορισμό προδιαγραφών που βοηθούν την ομαλή κυκλοφορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ασφάλεια. Οι προασπιστές της ασφαλείας είναι αυτοί οι φορείς, αυτοί οι οργανισμοί. Υποστηρίζουν αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε να επικρατεί, να έχει πρώτη θέση ασφάλεια. Βέβαια θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια στοιχεία αφορούν την ασφάλεια και θα διαβιβάζονται άμεσα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια στους οργανισμούς. Τελείωσε ο χρόνος. Ο κ. Λιμπεράτσκι για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αποψήφια Επίτροπε, ας αρχίσω πρώτα για το εμπάργκο. Υπάρχει, γίνεται λόγος για αποζημίωση για τους ε, αγρότες και τα λοιπά σε τέτοιες περιπτώσεις. Κανείς όμως δεν ε, μιλά για αποζημίωση των ε, μεταφορών. Και οι ζημίες ανέρχονται σε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Μπούλτς, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ονειρεύεται έναν Ευρωπαίο Υπουργό Μεταφορών. Τι σημαίνει βέβαια αυτό. Εσείς ως ε, επίτροπος μεταφορών πώς θα υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των ε, ε, εταιριών στο παγκόσμιο εμπορικό στερέωμα έπειτα. Υπάρχει και αυτό το όνειρο της σταθεροποίησης περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων για τις επιχειρήσεις. Βέβαια, Μ' άρεσε πάρα πολύ που άκουσα τις απόψεις σας. Δεν ξέρω όμως ποια θα είναι και η τελική συστασή σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να πω πως ε, είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί με το εμπάργκο. Το εμπάργκο από τη Ρωσία είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να το προβλέψεις σε στάδιο σχεδιασμού. Βέβαια, πιστεύω πως δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωστόσο, όντω δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, πρέπει να το συζητήσουμε και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει αρκετά. Όμως, το άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πώς δηλαδή οι ευρωπαϊκές ε, μεταφορές θα μπορούν να σταθούν στο παγκόσμιο εμπορικό γίγνεσθε. Πώς. Η Ευρώπη πρέπει να παραμένει ανοιχτή. Εάν θέλουμε να είμαστε ένας σημαντικός παίκτη παγκόσμια, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Εγώ θα υπερασπιστώ και θα πολεμήσω για την ε, δικαιοσύνη στον τομέα αυτό, για την αμοιβαιότητα των σχέσεων. Δεν γίνεται δηλαδή να δίνουμε συνέχεια και να μην παίρνουμε. Όμως εδώ μπορώ να σας πω ότι έχετε έναν ε, πάρα πολύ αξιόλογο προασπιστή των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Διότι έχω εντοπίσει κάποιους ε, τομείς ε, στους οποίους θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Οι αερομεταφορές για παράδειγμα. Υπάρχουν όλα, όλοι αυτοί οι σταθμοί τα αεροδρόμια στι ε, άκρε τη Ευρώπη, παρυφέ τη Ευρώπη, που θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να υπερασπιστούμε αυτού ε, του ε, σταθμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτό φαίνεται και στι μεταφορέ γενικότερα. Όμω, ναι, εγώ θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα τη Ευρώπη. Κύριε Αρναούτου. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Δεσμευθήκατε να επιδιώξετε την πολιτική φιλελευθερωποίηση σε όλους τους τομείς, κυρίως για τις μεταφορές. Πρέπει να ξεκινήσουν για θεσμικές συνομιλίες του τέταρτο πακέτο για τους σιδηρόδρομους. Και διατείνεστε ότι πάντα θα ζητάτε περισσότερο ανταγωνισμό στους σιδηροδρόμους για τη μεταφορά επιβατών, διότι λέτε η έλλειψη ανταγωνιστικότητας θα οδηγούσε σε υψηλές τιμές και μείωση της ποιότητας. Κυρία Επίτροπε, Είμαι Γάλλη εκπρόσωπος, Γαλλίδα εκπρόσωπος και δεν έχω πρόβλημα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ήταν πρόδρομος στις δημόσιες υπηρεσίες κυρίως για τα τρένα μεγάλης ταχύτητας και είναι πιο, τα πιο ασφαλή στον κόσμο. Και είναι δημόσιος τομέας σιδηρόδρομη. Στο μέλλον θα ακούτε τη φωνή εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης και κυρίως των Γάλλων που πέρσι απέρριψαν τον υπερβολικό φιλελευθερισμό και την τεχνοκρατία που πολύ συχνά ενσαρκώνεται στα μάτια του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία μου, θα μάθετε το παρελθόν που δείχνουν ότι η φιλελευθερωποίηση των σιδηροδρόμων μεταφράζεται πολύ συχνά με μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ασφαλείας των επιβατών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα το τέταρτο αυτό, η τέταρτη δέσμη μέτρων δεν αφορούν αποκλειστικά τα μέτρα την απελευθέρωση, φιλελευθεροποίηση, αλλά λειτουργικότητα, ασφάλεια, διαφάνεια και όταν μιλάμε για την επιχειρηματική πτυχή όπως προανέφερα οι χώρες δεν έχουν μία και μοναδική προσέγγιση. Το ξέρω πρέπει να αποφασίσουμε έναν κοινό τόπο και θα πολεμήσω για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, διαφαν... διαφάνεια. Να βλέπουμε πώς γίνονται οι κρατήσεις, ε, να υπάρχουν, ε, ναι, πώς καθορίζονται οι τιμές. Να μην υπάρχει αδιαφάνεια και να υπάρχει επιδότηση από μια υπηρεσία προς άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει σε κάποιο βαθμό κάθετη ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Θέλουμε να μην υπάρχει επιδότηση αδιαφανής. Αυτό δεν αφορά τη φιλελευθερωποίηση αυτή καθε αυτή, αυτό αφορά διαφάνεια. Θα πρέπει η προσέγγιση μας να εδράζεται επί του κόστους. Μιλάμε για χρηματοδότηση και επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είμαστε συνεπώς βέβαιοι σε τι επενδύουμε. Και άλλο θέμα. το επίπεδο της διαχείρισης και διοίκησης που είναι σημαντικό επίπεδο αφορά την ασφάλεια, τη διαφάνεια και καλύτερη παροχή υπηρεσιών και όχι τη φιλελευθεροποίηση. Είναι κάτι που θα είναι υποφελές και για τα σιδηροδρομικά συστήματα και επιβάτες πιβάτες. Evans, η κυρία Evans έχει το λόγο μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρατε πολλές φορές απόψε την ανάγκη για ουσιαστικές επενδύσεις στον χώρο των μεταφορών και για λόγους οικονομικούς και για λόγους ασφαλείας, για τουρισμό, περιβαλλοντος και Φυσικά αυτό θα γίνει και μέσω του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και μέσω της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη που είναι και το κέντρο της πολιτικής μας. Χρειάζονται όμως επενδύσεις και σε τομείς με ιδιαίτερα περιφερειακό χαρακτήρα και αναφερθήκατε λίγο σε αυτό. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία και είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της μεγάλης ανάγκης βελτίωσης των μεταφορών στις περιφέρειες. Και μάλιστα ιδιαίτερη σημασία έχουν οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Πώς λοιπόν εσείς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα λησμονηθούν αυτές οι περιοχές των μεταφορών. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει και τις ανάγκες ε, των, περιφερειακών, ε, των περιφερειών. Ε, υπάρχουν κάποια ταμεία τα οποία είναι τα διαρθρωτικά ταμεία συνοχής και είναι τουλάχιστον για τη δική μου χώρα από τις κυριότερες πηγές επενδύσεων. Φυσικά, υπάρχουν και ε, διάφοροι περιορισμοί στη χρήση αυτών των κονδυλίων, για παράδειγμα περιβαλλοντικοί ε, περιορισμοί. Κάτι άλλο το οποίο έχουμε συζητήσει είναι νέους ε, καινοτόμους μηχανισμούς οι οποίοι πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έτσι ώστε να μπορέσουν να ταπεξέλθουν στις ανάγκες των περιφερειών. Βέβαια είναι και στο χέρι των κρατών μελών να ψάξουν να βρουν αυτούς τους ε, μηχανισμούς και να βρουν τις επενδύσεις που χρειάζονται. Να σας αναφέρω και το παράδειγμα της Σλοβενίας, ήδη γίνονται κάποιες συζητήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο για την έβρεση αυτών των ε, πόρων. Επίσης διάβασα στους ε, Financial Times πρόσφατα ότι οι, συ, οι σιδηροδρομικές ε, εταιρείε μεταφορών ήδη προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ταμεία συνοχής. Δεν μπορώ δυστυχώς να σας προτείνω κάποια πιο καινοτόμο λύση αυτή τη στιγμή, όμως σίγουρα προτίθεμαι να την αναζητήσω και φυσικά ελπίζω στην ανταλλαγή βρέλτης των πρακτικών, διότι κάτι που μπορεί να λειτουργεί καλά σε μια περιοχή μπορεί να λειτουργήσει καλά και σε κάποια άλλη. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές καλές ιδέες στον τομέα αυτό και πρέπει να αξιοποιηθούν. Τάνια Γκοντζάλε Πένιας από την ΚΟΥ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Αποψήφια Επίτροπε, θα ρωτήσω εσάς το ίδιο πρότσα και τον κύριο Σεύκοβιτς και ελπίζω να μου δώσετε μία ε, πιο ξεκάθαρη και λεπτομερή απάντηση. Η στρατηγική της Ευρώπης 2020 έχει ως στόχο την πρόθεση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. Ωστόσο, παρατηρούμε μια ανεπαρκή συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριμένους ε, ε, τομείς, ιδιαίτερα στις μεταφορές που θεωρούν τους επενδυτές ανώτερους από τους ίδιους τους κατανάλωτες, τους χρήστες για παράδειγμα το έχουμε δει αυτό να γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχουν μετά κάποια ε, οδικές αρτηρίες, κάποια διόδια που πρέπει να τα αναλάβουν οι κυβερνήσεις. Μετά κάποιοι δρόμοι που, αυτοκινητόδρομοι που πρέπει να ε, μπορούν να σηκώσουν ε, φορτίο φορτηγών. Υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί. Πώς εσείς λοιπόν μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η πολιτική των μεταφορών θα είναι σχεδιασμένη από, τους, ε, από ανθρώπους για ανθρώπους, για τους χρήστες και θα έχουν κύριο μέλημά τους το καλό των χρηστών παρά το να υπακούν τυφλά τα συμφέροντα των επενδυτών. Και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Uh, Αλλά έχουν τεθεί κάποια προγράμματα από το Κοινοβούλιο, το εμπιστεύομαι και θα εξασφαλίσω την εφαρμογή τους. Όλα έχουν σχεδιαστεί στα πλαίσια του ΣΕΦ. Ακούω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω. Κατανοώ ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Κυρίως όσον αφορά τον κόσμο. Έχω πιστεί προετοιμαζόμενοι για την ακρόαση ότι όλες αυτές οι επενδύσεις για τις υποδομές που έχουν ευρύτερο σκοπό θέλουν να υπάρχει μια ομαλή κυκλοφορία στην Ευρώπη αν το πετύχουν δεν θα είναι κάτι εποφελές μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και οι επιβάτες θα επωφεληθούν κατά πολύ σε κάθε βήμα σε κάθε τι που κάνουμε έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να ακολουθούμε πράσινη προσέγγιση και πράσινο θεματολόγιο. Τα τελευταία δέκα χρόνια είδα ότι όλα τα προγράμματα εφαρμόστηκαν σε τεχνικό επίπεδο, οργανωτικό επίπεδο, δημιουργήθηκαν επιχειρηματικά μοντέλα και όλες αυτές οι προσπάθειες ακολουθούν μια πράσινη κατεύθυνση. Αν πέτυχαν όλα το στόχο τους, όχι, διότι είναι άνθρωποι πίσω από τις προσπάθειες έχουμε δυνατότητα βελτίωσης. Εν γέννη όμως ακολουθούμε σωστή κατεύθυνση. Επιτυγχάνουμε στόχους που κανείς άλλος στον κόσμο δεν πετυχαίνει και ελπίζω ότι θα μπορέσω αυτό να το εξάγω σαν έννοια. Μόνο αν εξάγουμε αυτές τις έννοιες θα μπορέσουμε να τις ζήσουμε πραγματικά. Δεν μπορεί να είναι απομονωμένο η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να διαβιβάσει, να στενιστούν και άλλοι τις δεσμεύσεις. Ματέις Φων Βίτεμπουργκ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για ένα θέμα που θα θέσω στα Ολλανδικά για το χρόνο ανάπαυσης. Ίσως είναι και επί και αυτή την ώρα. Λοιπόν, χρόνο ανάπαυσης στον οδικό τομέα, των οδικών μεταφορών. Λοιπόν, Ολλανδικά. Λοιπόν, για να πετύχουμε σωστή προσέγγιση για τις οδικές μεταφορές, για το σωστό ανταγωνισμό, θα πρέπει να Υπάρχει ομοιομορφία όσον αφορά την νομοθεσία που αφορά τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα αυτού των κανόνων. Στη Γαλλία ο χρόνος ανάπαυσης στο φορτηγό όταν κοιμάται ο οδηγό στο φορτηγό δεν θεωρείται ότι είναι επίσημος χρόνος ανάπαυσης στη Γαλλία και μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις μέχρι 30.000 ευρώ και φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο. Όταν κανείς κοιμάται, ο οδηγός κοιμάται μέσα στο θάλαμο του οδήγησης. Σε άλλες χώρες δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Σαν επίτροπος, τι θα κάνετε για αυτό το θέμα Πώς θα φροντίσετε το ώστε η εφαρμογή των κανόνων για τον χρόνο ανάπαυσης να είναι πιο ομοιόμορφη και να γίνονται σεβαστοί καλύτερα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Απάντηση. Με ενημέρωσαν για αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι δεν γνωρίζω πώς προήλθε ε, θα πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα πώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου όσον αφορά το θέμα αυτό και την επιβολή των κανόνων. Χρειάζομαι λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται να κατανοήσω γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα αλλά θα ήθελα να συμφωνήσουμε επί βασικών κανόνων κοινών ποιοι θα είναι στο μέλλον. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι κανόνες. Θα δούμε ποιες είναι οι ανάγκες. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και συναρτήσει αυτόν θα κινηθώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γνωρίζω το πρόβλημα, αλλά δεν γνωρίζω αρκετά ούτως ώστε να σας δώσω μια λύση. Και λυπούμε πολύ γι' αυτό. Ρομπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ πολύ, Μίχαλ. Κύρια Πούλτ, Μιλάτε για την αμοιβαιότητα και συμφωνώ μαζί σας όταν έχουμε τις ε, ε, θέμα της διακριτικής μεταχείρισης. Ε, τι πιστεύετε για το θέμα των, των υπερπτήσεων πάνω από την Ουκρανία... για τις υπεσιβηρικές υπεπτήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αντιδράσει με αμοιβαιότητα εάν ε, οι Ρώσοι ε, επιδοτούν τις δικές τους πτήσεις. Ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι τα τέλη είναι παράνομα για αυτές τις ε, πτήσεις. Ε, τα τέλη είναι παράνομο, όχι πτήσεις. Ε, πρέπει να είμαστε όμως πάρα πολύ προσεκτικοί διότι σε αυτήν την τεταμένη πολιτική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει με τη Ρωσία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Από όσο ξέρω τους Ρώσους δεν πρέπει να εξαφανιστούν αυτά τα ζητήματα. Η Ρωσία από ό,τι κατάλαβα αποφάσισε να καταργήσει αυτά τα τέλη με την προσχώρηση στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πολλοί συναδελφοί μου είπαν ότι θα λύσουν το ζήτημα. Ε, αν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα τα καταφέρω, δεν μπορώ να το υποσχεθώ, αλλά θα χρειαστεί να με βοηθήσετε για να τα καταφέρω. Είναι μεγάλη πρόκληση και δύσκολο να πιέσει κανείς τη Ρωσία να κάνει κάτι που δεν θέλει. Πρέπει να δούμε ποια εργαλεία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να το πετύχουμε. Πάντως, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια και αν με επιλέξετε, ευελπιστώ να μπορέσω και να λύσω το ζήτημα. το Κύρκος. Συγχαρητήρια κυρία Μπόλτς και σας εύχομαι καλή επιτυχία και για σας αλλά και για την Επιτροπή μας. Η ερώτησή μας τώρα, πώς θα αξιολογούσατε το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα, τι προσδοκίες θα είχατε από το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και εκτός από το πακέτο, τι χρειάζεται η Ευρώπη ακόμα για να βελτιώσει το σύστημά της. Ευχαριστώ. As Όπως είπαμε ήδη, το, είναι πολύ σημαντικό το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και σας είπα ότι δεν θέλω ένα πέμπτο. Ε, παλέψουμε λοιπόν για το τέταρτο. Τώρα συμβαίνει αυτό και το τεχνικό του κομμάτι είναι ε, σημαντικό διότι ε, Υπό τον τίτλο του Refit, χιλιάδες διαφορετικοί κανόνες και νομοθετήματα θα ενοποιηθούν, θα συγχωνευτούν, θα απλουστευτεί η διαδικασία και έτσι ε, θα λειτουργεί ομαλά και χωρίς ε, διακοπές το δίκτυο μεταφορών στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το όραμά μας. Θέλουμε αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος για το δίκτυο μεταφορών. Θέλουμε ε, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις μας να έχουν στη διάθεσή τους ένα αποτελεσματικό δίκτυο μεταφορών. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Στο επιχειρησιακό και στο τεχνικό κομμάτι τα επιμέρους στοιχεία είναι μικρά-μικρά βηματάκια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα υπάρξουν πολλά στοιχεία λοιπόν μέσα στο τέταρτο συνδρομικό πακέτο που θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια του δικτύου. Τώρα η διατροπικότητα και η διελειτουργικότητα είναι δύο πολύ σημαντικές συνιστώσεις. θα επιτρέψουν καλύτερη εφαρμογή των δεσμεύσεων μας, των οικολογικών μας δεσμεύσεων, αλλά θα προστατεύσουν επίσης και τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά όχι μόνο, με θεαματικό τρόπο θα ε, βελτιωθούν οι συνθήκες ε, με τις οποίες, υπό τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά μου, διότι κουράζομαι και με καταλείπουν σιγά σιγά. Ελπίζω πως σε συνεργασία μαζί μας και με το Συμβούλιο θα επιτύχουμε όλοι ε, να υλοποιήσουμε το τέταρτο συνδρομικό πακέτο. Ευχαριστούμε κυρία Λουκασιέμσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αποτιμάτε την κατάσταση ως προς το καμποτάζ σήμερα. Τι θα κάνετε για να αναπτυχθεί το δυναμικό αυτού του τομέα θα επιδιώξετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θα επιθεωρήσετε την εφαρμογή των κανόνων. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τους φορείς που έχασαν χρήματα λόγω του εμπάργου που επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία. Απάντηση. Πιστεύω πως το καμποτάζ είναι ένα πρόσφορο μέτρο για να βελτιστοποιήσουμε την δυναμικότητα των μεταφορών που έχουμε στη διάθεσή μας ταυτόχρονα είναι και μία μικρή συμβολή στην πράσινη ατζέντα για την Ευρώπη. Όπως σας είπα, έχω λειτουργήσει στον τομέα της ε, υλικοτεχνικής υποστήριξης όχι άμεσα, αλλά πελάτες μου εξαρτώνταν από τα μέτρα για την υλικοτεχνική στήριξη και ο μεγαλύτερος φόβος τους ήταν να ε, είναι ε, άδεια τα, τα φορτηγά στους δρόμους. Οπότε έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μετακινούνται φορτωμένα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Να μιλήσουμε με αυτούς που άμεσα συμμετέχουν, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς αυτούς. Η νομοθεσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει να εξυπηρετεί τους χρήστες. Αυτή θα είναι η στάση που θα τηρήσω για νέες υπηρεσίες ή νέα μοντέλα που θα προκύψουν, νέες ιδέες που θα προκύψουν, διότι πέρα από την βελτίωση αυτών που ήδη έχουμε, ένας βασικός μας στόχος είναι επί τη βάση των νέων δυναμικών και των νέων αναγκών μας να επιζητούμε διαρκώς νέες λύσεις. Αυτές χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου ενιαίου χώρου μεταφορών παραμένοντας ανταγωνιστική και να μην ξεχνάμε ποτέ τα βασικά στοιχεία όπως η οδική ασφάλεια. Αυτό δεν συνδέεται άμεσα με το καμποτάζ, το ξέρω, αλλά είδω αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστούμε, Μπάς Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι, κυρία Μπολτσα. ε, μας εξηγήσατε ότι αγαπάτε όλους τους τρόπους μεταφορών. Αυτό το κατάλαβα από τις απαντήσεις σας μέχρι στιγμής. Ε, αν δούμε όμως ε, την τιμολόγηση των τρόπων μεταφοράς βλέπουμε διαφορές. Ε, η αεροπορία δεν ήταν μέρος οποιοδήποτε συστήματος τιμολόγησης και δεν ήταν ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών σε σχέση με τις σιδηροδρομικές. Τι θα κάνετε λοιπόν για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα ανταγωνισμού που προς το παρόν ευνοεί την αεροπορία εις βάρος των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, μετά το 2016 θα μπορούσε να είναι τμήμα του ETS, ε, του συστήματος ε, εμπορίας ρήπων ε, όταν ευελπιστούμε θα επικρατήσει και ένα παγκόσμιο τέτοιο σύστημα ρύθμισης των δικαιωμάτων εκπομπών. Απάντηση. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ευρωπαϊκές αεροπαρικές εταιρείες, έτσι δεν είναι. Εγώ θα έτεινα να θέσω το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο και να το συζητήσουμε στα πλαίσια ενός ε, πολυμερούς διεθνούς οργανισμού. Αυτό το ζήτημα απορρέει από την ιστορική εξέλιξη. Η αεροπορία είναι στη θέση που είναι λόγω των πολιτών εξελίξεων στον τομέα αυτό. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι το 2016 η αεροπορία θα μπει στο, φάγκος, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων. Θα ήταν υπερβολικό να το υποσχεθώ. Η αεροπορία σίγουρο είναι πως πρέπει να εξελιχθεί, να αρχίσει ο διάλογος για αυτό το ζήτημα και θα χρειαστώ την υποστήριξή σας. Από κοινού με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις και να υποβάλουμε προτάσεις. Σε συνεργασία μαζί σας όμως θα βρούμε ε, το δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Δεν μπορώ μέχρι το 2016 να σας προσχεθώ θα μπει στο ETS, αεροπορία και συμφωνώ με αυτό που είπατε ε, για το χάσμα ότι δεν, είναι, ε, δεν λειτουργούν σε ισότιμη βάση οι διάφοροι τρόποι μεταφορά περώτηση. Ε, Έχω 25 δευτερόλεπτα ακόμη, λέει ο κύριος Έκχατ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι βάσει της νομοθεσίας, ότι αν το 2016 δεν υπάρξει παγκόσμια συμφωνία, η αεροπορία θα ενταχθεί στο ETS. Το έχει πάρει απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντηση. Ε, θα φροντίσουν να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Πολύ ωραία. Μαλτέζα από την Κούρ. Περιμένοντα να υιοθετηθεί να εγκριθεί το τέταρτο πακέτο για του ιδεοδρόμου με προδιαγραφέ ασφαλεία, θέλω να ρωτήσω την Επίτροπο αν θεωρεί σκόπιμο να παρέμβει επί κάποιων των θεμάτων. Ένα από αυτά είναι φορτιστεί Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδεοδρόμων για την ασφάλεια να δράσει για να μειωθεί η ταχύτητα των τρένων αμέσως όταν μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, όταν περνάνε από αστικέ περιοχές. Στην Ιταλία είχαμε τραγωδία. 34 νεκροί του Βιαρέτζο. Ήταν ένα τύχημα που δυστυχώς θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στην Ένωση. Δεύτερο κατεπήγον θέμα. Ε, λοιπόν, ε, ε, χρησιμοποιώντας το GSM, που χρησιμοποιούν τα τρένα και χρησιμοποιούνται σε χερσαίες. Χρησιμοποιούν και ιδιωτικοί φορεί των τηλεπικοινωνιών κάποιες συχνότητες και μπορεί να δημιουργηθεί παρεμβολή επικίνδυνη όπως το Βέλγιο το Φεβρουάριο του 2013. Η Ελβετία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέλυσε αυτή τη σύγκρουση συχνοτήτων υπέρ της ασφαλείας των πολιτών. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει κάτι παρόμοιο. Απάντηση. Καταρχάς να προσπαθήσω να απαντήσω στο πρώτο σας ερώτημα εάν θα προχωρούσα δεν θα υποστήριζα τέτοιες δράσεις θα ρωτήσω εσάς το Κοινοβούλιο για να προωθήσουμε το πακέτο ταχύτερο δυνατόν ε, εμπεριέχει πολλά ωφέλη δεν θέλουμε να προωθήσουμε μόνο μερικά κομμάτια του πακέτου για να μην διαλυθεί το πακέτο. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ό,τι δυνατότητες έχουμε για να εγκριθεί το πλήρες πακέτο. Με ενημέρωσαν για τα προβλήματα που υπάρχουν και κάποια τα τυχήματα που συνέβησαν ε, λόγω της κακής διαχείρισης των δικτύων και των σημείων διασύνδεσης. Ελπίζω ότι με το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας που δεν θα έχει εμπόδια, θα λύσουμε τα προβλήματα. Δεν θα υπάρξουν ξανά τέτοια προβλήματα. Είδα την εικόνα, είναι απίστευτο. Είναι φρικτό όταν βλέπει κανείς ότι υπάρχουν τέσσερα ή πέντε διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και πρέπει κανείς να τα διαχειριστεί και να αντιδράσει. Είναι απαράδεκτο αυτό για τη σύγχρονη κοινωνία. Κυρίως όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής. Αντί να βρούμε μερικές λύσεις, εγώ θα έλεγα να προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε συστημικοί στην προσέγγιση μας. Να αντιμετωπίσουμε συστηματικό τρόπο τις προκλήσεις. Να βρούμε γενικές οριστικές λύσεις που μακροπρόθεσμα θα εμποδίσουν να συμβούν και άλλα τέτοια τυχήματα. Παύλ Τιλίτσκα. Καλησπέρα. Ε, ε, καλωσορίσατε ο Μάρκος Σιφκοβίτς, ε, πολύ καλός μου φίλος. Ε, επίσης ε, σας καλωσόρισε. Νομίζω ότι αξίζει ενθάρρυνση όποιος πρέπει να υποστεί μια τέτοια ακρόαση. Και πάλι αποφάσισε ο Πρόεδρος να ανακατανείμει τα χαρτοφυλάκια Είστε πάντως πάρα πολύ συγκεκριμένε απαντήσει που δίνετε και είχατε μόνο πέντε ημέρες στη διάθεσή σας για να προετοιμαστείτε και το εκτιμώ, εκτιμώ την προσπάθεια που κάνατε παρότι δεν με ικανοποίησαν οι, όλες οι απαντήσεις που δώσατε. Κατά τη γνώμη μου, όπως είπε ο κύριος Ζήλε, δεν προωθήσατε παρακώ στην αρχή του use it or lose it, χρησιμοποιήστε εδώ ή χάστε το. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει επαρκής απορρόφηση των κονδυλίων θα γίνεται ανακατανομή. Πρέπει να το ξανασκεφτείτε ίσως και να μου απαντήσετε ότι για να είστε αποτελεσματικοί και να είναι αποτελεσματική η απορρόφηση θα πρέπει να υπάρχει η απειλή της ανακατανομής των κονδυλίων. Στη συνέχεια για το εξωτερικό κόστος μιλήσατε για ένα όραμα που έχετε και Τώρα ψάχνετε ένα μηχανισμό που θα βασίζεται ε, στον υπολογισμό του κόστους επαρκή. Νομίζετε μιλήσαμε για τη Γερμανία, ε, η Γερμανία μίλησε ε, ο Γάλλος Υπουργός για τη φορολόγηση των φορτηγών. Εσείς θα μπορούσατε να είσαστε λίγο πιο φιλόδοξοι σε ένα λεπτό. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να σας απαντήσω διμερώς. Ας προσπαθήσω το αχύτερο δυνατόν να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Use it or lose it, χρησιμοποιήστε τα ή χάστε τα. Πιστεύω ότι είναι πολύ ε, καλή αυτή η αρχή, καλη αυτη η αρχη μιλω εξ πείρας, έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το είδα ε, στη χώρα μου, χρειαζόμαστε όμως και τα κατάλληλα εργαλεία γι' αυτό. Πώς μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή, αν είναι σαφής ο μηχανισμός, να λέει, πολύ ωραία, υποβάλλετε και σχεδιάζετε το πρόγραμμά σας, εάν δεν ε, πληρείτε τις υποχρεώσεις, τότε χάνετε τα λεφτά και μπαίνουν σε ένα κοινό ταμείο. Και όλες οι επιλέξιμες χώρες για το Ταμείο Συνοχής μπορούν να υποβάλουν τη δική τους προσφορά και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για ένα άλλο πρόγραμμα. Να δοθούν τα χρήματα και να ενθαρρύνονται αυτοί που μπορούν να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και να το μερούνται οι υπόλοιποι. Ρόμπερτ Τζίλε. Μετά τον κύριο Τελισκάτς με αυτή τη δύσκολη ερώτηση δεν χρειάζεται να... Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Μπορεί να κάνει ίσως ένα διαλυματάκι, η κυρία Μπούλς για να ξεκουραστεί. Βάνο Εδώ πίσω. Επίτροπε, εγώ είμαι ο τελευταίος ομιλητής από τους, ε, την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Νομίζω ότι ε, Ε, θα ε, ήταν σκόπιμο να σας μιλήσω για το διαγωνισμό ταλέντων X-Factor. Όταν έρχονται οι τραγουδιστές την πρώτη φορά η κριτική επιτροπή μετά από 20 δευτερόλεπτα μπορεί να πει ότι ναι, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί ξέρουν να τραγουδήσουν. Ε, δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είχατε τέσσερις ημέρες στη διάθεσή σας και εγώ Τέσσερις μήνες χρειάστηκα για να ενημερώθω, για να πρέπει να λάβω ε, ως αντιπρόεδρος. Ίσως καταφέρετε κάποια στιγμή σύντομα στο μέλλον να, να τραγουδήσετε με ικανοποιητικό τρόπο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει η Επιτροπή μας. Ε, λοιπόν, στον τομέα των μεταφορών είναι πολλά τα οργανωτικά και υπερβαλλοντικά ζητήματα και όταν δούμε στα Βαλκάνια και στι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες ε, πόση μεγάλη καθυστέρηση υπάρχει, συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο θα είναι να αναλυθούν συγκεκριμένα μέτρα. Εσείς έχετε πρόθεση σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο να δώσετε μια νέα όθηση ε, στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Πιστεύω ότι για το επόμενο ζήτημα θα με υποστηρίξει ο κύριος Κράμερ. Ξέρω ότι επειδή η Προεδρεύη δεν δικαιούται να κάνει ερωτήσεις, πρόκειται για την ποδηλασία. Ο ποδηλατικός τουρισμός, ε, υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι για αυτό. Ε, ένα λεπτό θα σας δώσω παρότι θα ήθελα δέκα για την ενδιαφέρον το ζήτημα. Απάντηση θα προσπαθήσω να δω ε, ποιε ε, είναι οι προτεραιότητε και η ασφάλεια είναι μια ύψιστη προτεραιότητα. Οτιδήποτε έχει ε, να κάνει με την ασφάλεια πρέπει να με εφαρμοστεί πρώτο. Όμω, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η δεύτερη ερώτηση, επιτρέψτε μου να την απαντήσω πρώτη, διότι είμαι ένθερμη ποδηλάτρια και αν πάτε στην ε, Σλοβενία θα δείτε πάρα πολλέ φορέ του υπουργού να φεύγουν από τι συνεδριάσει των συμβουλίων με πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Όμω, εγώ παίρνω το ποδηλατάκι μου. Πραγματικά το λατρεύω το ποδήλατο. Και τα ταμεία συνοχή και τα διαθερωτικά ταμεία έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για την ε, ποδηλασία και του ποδηλάτε ε, στη χώρα μου. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει με πάρα πολύ καλό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ε, ελπίζω αυτή η κουλτούρα τη ποδηλασία να ενσωματωθεί σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βόζεμπεργκ έχει το λόγο ω τελευταία μιλήτρια για, τους για το ΕΛΚ. Κυρία να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι η τελευταία ομιλήτρια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και πραγματικά να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι σε ένα απαιτητικό χαρτοφυλάκιο ενημερωθήκατε τόσο γρήγορα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και οι απαντήσεις σας ήταν πλήρεις και τεκμηριωμένες. Δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω για τα λιμάνια, με το δεδομένο ότι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός οικονομικός μοχλός είναι, πόσο συμβάλλουν στην οικονομία της Ευρώπης και πώς το γεγονός ότι το 90% του ευρωπαϊκού εμπορίου διακινείται στη θάλασσα, τους δίνει μια αξία η οποία πρέπει και να θεσμοθετηθεί σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που έχει προτείνει νέο η Επιτροπή και αυτό στοχεύει ουσιαστικά σε δύο άξονες. Αφενός μεν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και περαιτέρω στο γεγονός ότι πρέπει πραγματικά να διασφαλιστεί η διαφάνεια που αφορά στη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Έχετε όμως υπόψη σας ότι υπάρχουν ισχυρές επιφυλάξεις και αντιδράσεις από κάποια κράτη-μέλη, από κάποιους φορείς, καθώς επίσης και σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή σε αυτή την κατεύθυνση του νομοθετικού πλαισίου που έχει προτείνει η Επιτροπή, ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε προκειμένου ε, με το δεδομένο αυτών των επιφυλάξεων στις οποίες αναφέρθηκα να αρθούν και να μπορέσει να προωθηθεί, να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο νόμου που θα προταθεί από την Επιτροπή. Και επίσης μια τελευταία ερώτηση που αν θέλετε έχει και ένα θεμητά ιδιωτελές πρόσημο, εθνικό πρόσημο για μένα γιατί προέρχομαι από την Ελλάδα που είναι νησιωτική χώρα και με ενδιαφέρει κατά πόσον στοχεύετε να συμβάλλετε στην περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λιμένων σε ό,τι αφορά σε νησιά και σε απομεμακρυσμένες περιοχές. Ειδικά στη χώρα μου υπάρχει αυτό το πρόβλημα και βέβαια με ευχαριστεί το γεγονός εφόσον αναλάβετε ότι θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας και σε αυτές τις κατευθύνσεις. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, ε, τα λιμάνια όντως είναι μέρος του θεματολογίου του ΣΕΦ. Και όπως προείπα, θα ακολουθήσω πιστά το θεματολόγιο. Γι' αυτό λοιπόν και ε, θα ακολουθήσω και τα όσα προβλέπει για τη χρηματοδότηση των λιμένων. Είναι, ε, υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ε, περαιτέρω χρηματοδότηση και πρέπει να δούμε τους υφιστάμενους ε, μηχανισμούς. Αλλά αυτό θα το δούμε και μακροπρόθεσμα. Είναι όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επεκταθώ αυτή τη στιγμή σε τόσο λίγο χρόνο. Όμω, όντω υπάρχουν οι προκλήσει ε, που αντιμετωπίζουμε από την Κίνα και πρέπει να ε, τι ε, λύσουμε. Μετά, με ρωτήσετε για τα ελληνικά νησιά. Θα ήταν καταπληκτικό μπορούσα να σας κάνω υποσχέσεις τώρα, όμως δυστυχώς δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας κάνω κάποια υπόσχεση. Οι εξελίξεις θα συνδεθούν και με το θεματολόγιο της επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό πιστεύω πως μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τα λιμάνια ελκυστικά για τους επενδυτές. Αυτή δεν ήταν μόνο η τελευταία ερώτηση για το ΕΛΚ, λέει ο πρόεδρος, αλλά και η τελευταία ερώτηση από την Επιτροπή Μεταφορών. Τώρα έχετε τη δυνατότητα για πέντε λεπτά να συνοψίσετε αυτά που είπατε και έχετε αμέσως.